Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει στο δεύτερο τμήμα της ακροασής μας που έχει να κάνει με τις περιφερειακές αλληλευτικές οργανώσεις. Θα ξεκινήσουμε στην ώρα μας, γιατί μετά δεν θα προλάβουμε για την τρίτη θεματική ενότητα να εξαντλήσουμε το θέμα μας. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως. Περιμένω βέβαια να δω να μπαίνουν και άλλοι ευρωβουλευτές για να ακούσουν για αυτό το θέμα που είναι τόσο ζωτική σημασία στο Κοινοβούλιο αυτή την εποχή, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου εννοείται. Έχουμε τρεις που θα πάρουν το λόγο σε αυτή τη θεματική ενότητα και που θα μιλήσουν 10 λεπτά ο καθένας. Και μετά θα έχουμε, όπως και σήμερα το πρωί, 50 λεπτά περίπου για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, θα πάρει το λόγο η κυρία Πηγιαρές, η οποία είναι υπεύθυνη του τμήματος ε, της Διεθνούς Επιτροπής για την διατήρηση των τονοειδών στον Ατλαντικό. Είναι υπεύθυνη και για το κοινογραφικό κέντρο της Ισπανίας. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας αυτή. Σας δίνουμε το λόγο ευθύ αμέσω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το ICAT που σημαίνει International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna στα αγγλικά. Είναι μια περιφερειακή οργάνωση αλίας y <clears throat> Υπάρχουν από το 1967 με αρχική ισχύ το 1969. Στόχος οργάνωσής μας ήταν να προστατεύσουμε τους σπόρους του Ατλαντικού που είναι βασικοί για την διατροφή. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε συμφωνία δύο φορές. Οι αρμοδιότητες είναι τα τονοειδή και τα συναφή είδη και ο χώρος που δρούμε είναι ο Ατλαντικός ωκεανός αλλά και οι γειτονικέ θάλασσες. Έχουμε 48 συμβαλόμενα μέρη με 98% των, ε, του συνόλου των αλλιευμάτων των ειδών και συναφών ειδών. Έχουμε διάφορα όργανα, όπως είναι η μόνιμη Επιτροπή για τα Δημοσιονομικά και τη Δίκηση. Έχουμε τέσσερις επιτροπές επίσης με ειδικέ ομάδες αναείδος. Έχουμε τη μόνιμη Επιτροπή για την έρευνα και τις στατιστικές που καλύπτει ε, διάφορα είδη. Και ασχολείται και με τις στατιστικές επίσης. Επίσης έχουμε και μια επιτροπή για τα διαχειριστικά μέτρα και μια ομάδα μόνιμη εργασίας. Έχουμε τη γραμματεία η οποία έχει ως ρόλο να στηρίξει τους διάφορους τομείς και τα διάφορα σώματα της Επιτροπής αυτής. Γίνονται αξιολογήσεις των αποθεμάτων των ειδών, υπάρχουν και προγράμματα ερευνητικά και παρακολουθούμε θέματα που έχουν να κάνουν με το οικοσύστημα. Αξιολόγηση επιστημονική επίσης, όπου βοηθάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δικό της έργο και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε ζητήματα τα οποία βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τα νεστευτικά είδη των τόνο και οι αξιολογήσεις που γίνονται από την Επιτροπή μας βασίζονται σε δεδομένα που έχουμε από τις ελευτικές ζώνες. Η διαθεσιμότητα των ε, στοιχείων λοιπόν αποτελούν πολύ βασικό θέμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αξιολογήσεις. Ε, μια πολύ βασική αρχή Τη οργάνωσή μα και των διαφόρων επιτροπών μα είναι διαφάνεια. Γι' αυτό και θέλουμε να συμμετέχουν όλα τα διαφερόμενα μέρη στι ομάδε εργασίας. Δεν συμμετέχουν λοιπόν μόνο τα συμβαλόμενα μέρη, αλλά και παρατηρητές και έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, είναι στη διάθεση του κοινού. Έχουμε δραστηριότητε όσον αφορά τη διαχείριση των παρών και εκεί τα συμφελόμενα μέρη είναι υποχρεωμένα να δίνουν στοιχεία και για ονομαστικά αλλιεύματα και για λεπτομέρειες ανα είδος, πόρους, ανα μέγεθος αλλιευτικού σκάφους και άλλα στοιχεία. Ετησίως μάλιστα. Ένα πολύ βασικό θέμα είναι πώς να εμφανίσουμε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εύκολα αυτός που παίρνει την απόφαση της διαχείρισης των ειδών, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση. Στην πρώτη κοινή συνεδρίαση των Περιφερειακών Οργανώσεων αλία των Ειδών τέθηκε αυτό το θέμα και καταλήξαμε σε μια συμφωνία για μια γραφική απεικόνηση ανάλογα με την βιομάσα και το, την παραγωγή των ειδών και το άλλο ανάλογα με τις επιπτώσεις που έχει η αλία. Και οι δύο παράμετροι αυτοί έχουν να κάνουν με τους στόχους της σύμβασης. Ο τρόπος αυτός απεικόνησης είναι ένα τετράγωνο όπου αναφέρονται οι στόχοι από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά του τετραγώνου αναφέρονται τα αποτελέσματα της υπεραλίευσης. Βάσει λοιπόν αυτού του σχεδίου, αυτής της απεικόνησης, έχουμε δύο τρόπους να παρουσιάζουμε τις αξιολογήσεις μας. Το ένα είναι ο πίνακα Scope, που δείχνει ποια είναι η κατάσταση των ειδών. Βλέπετε εδώ πέρα από το κόκκινο μέχρι το πράσινο ε, τετραγωνάκι και το κόμπα Track που δείχνει τη διαδρομή. Επίση, καταλήγουμε και σε έναν πίνακα συνοπτικό που δείχνει, μπορεί κανείς πολύ εύκολα να δει ποια είναι η κατάσταση των αποθεμάτων ανάλογα με τη διαχείριση. Στη συνέχεια, τις ε, πληροφορίες τις εμφανίζουμε από μορφή συστάσεων διαχείρισης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη δεύτερη κοινή συνάντηση που είχαμε οι περιφερειακές οργανώσεις αλίας των ειδών, σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση λοιπόν αναπτύχθηκε ο λεγόμενος COB ε, Matrix που είναι ένας πίνακας που βοηθάει για τη λήψη αποφάσεων. Και εκεί αναφέρονται τα μέτρα διαχείρισης που θα έπρεπε να ληφθούν για να πετύχουμε τους στόχους μας βάσει των, του νόμου των πιθανότητων βέβαια για μια συγκεκριμένη περίοδο. Εδώ λοιπόν μπαίνουν τα επίπεδα και τα ανώτατα επιτρεπόμενα λιεύματα. Τώρα, βάσει των άρθρων 8 και 9 της Σύμβασης λειτουργούμε βασιζόμενες επιστημονικές αξιολογήσεις προκειμένου να προστατεύσουμε τους στόχους της Σύμβασης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε υιοθετήσει πάνω από 10 συστάσεις ετησίως και ο μεγαλύτερος αριθμός συστάσεων έχει να κάνει σήμερα με τη συμμόρφωση στους κανόνες. Πρόκειται για συλλογή πληροφοριών που μας βοηθούν να αξιολογήσουμε την συμμόρφωση προς τους κανόνες με κατάλογο, με σκάφη άνω των 20 μέτρων, όσον αφορά καταλόγους επίσης σκαφών που κάνουν παράνομη αλίευση και άλλες πληροφορίες κατά εξάμεινο ανάλογα με τα είδη που προστατεύονται εκθέσεις όσον αφορά τις απαγορευμένες περιοχές, δηλαδή απαγόρευση αλίευσης για ένα χρονικό διάστημα, για τις αστηριότητες στα λιμάνια κλπ. Επιπλέον τώρα από τα γενικά μέτρα για τον ε, κόκκινο τόνο έχουμε μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες με καταλόγους και ειδικά μητρώα όσον αφορά τον, ε, τον αυτόν, τον μικρόπτερο για την πάχυνση επίσης ε, των ε, ψαριών και άλλες πληροφορίες επίσης μας ενδιαφέρουν, όπως είναι οι ποσότητες που βρίσκονται τόνο, δηλαδή που βρίσκονται σε κλουβιά για πάχυνση, ή για σκάφη άνω των 15 μέτρων, δηλώσεις όσον αφορά τις, ε, την αλίευση που γίνεται με παγίδες, με νέδρες για τόνο και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το είδο αυτό. Το 2010 μάλιστα ξεκίνησε και ένα περιφερειακό πρόγραμμα παρατήρησης για τον μικρότερο τόνο όσον αφορά σκάφη με γρηγρή, με γρήπο και επίσης για την ε, πάχυνση μέσα σε κλουβιά. Επιπλέον, συμμετέχουμε στο κοινό πρόγραμμα ελέγχων και εποπτείας. Πρόσφατα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε διάφορες προκλήσεις με δράσεις από τις οποίες θα σας αναφέρω την ε, μεταρρύθμιση της δραστηριότητας από κοινού με διάφορες περιφερειακές οργανώσεις των ειδών στο Κόμπε. Είχαμε τρεις εμπειρογνώμονες για τη διαχείριση επιστημονικούς επίσης με αποτελέσματα τα οποία συμπεριλήφθηκαν στα διάφορα επικουρικά όργανα, για παράδειγμα στην ομάδα εργασίας που έχει ο οργανισμός μας. Όσον αφορά τώρα την αρχή της πρόληψης, η ΚΑΤ δημιούργησε μια ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό, για την πρόληψη δηλαδή, ήδη από το 1998-1999 και στη συνέχεια έγινε μια κοινή συνεδρίαση η ΚΑΤ ΚΑΝΕΤ με ομάδα εργασίας για την ε, μέτρηση, όπου προσπάθησε μονοθεματικά να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Για το οικοσύστημα τώρα και τη διαχείρισή του. Η ΚΑΤ δημιούργησε μια υποεπιτροπή οικοσυστήματος, η οποία αξιολόγησε τις επιπτώσεις ε, της αλίευσης στα Και επίσης κάναμε και αξιολογήσεις για τα αποθέματα της ε, Σαρδέλας και άλλων. Όσον αφορά τώρα την ε, στήριξη χωρών υποανάπτυξη, το 2003 η ΚΑΚ δημιούργησε μια βάση δεδομένων που χρησιμεύσε για το πρόγραμμα βελτίωσης των δεδομένων διαχείρισης που λειτουργεί από το 1994. Το 2008 είχαμε και χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κονδύλια αυτά απευθύνονται για να, διευκολυνθούν, να διευκολυνθεί μάλλον η συλλογή επιστημονικών δεδομένων, όπως επίσης για να δημιουργούνται εργαστήρια, ενημέρωση κλπ. Όσον αφορά τα ερευνητικά προγράμματα τώρα που ζητάει η ΚΑΤΑ συνεχώς, φέτος ξεκίνησε ένα πρόγραμμα όσον αφορά τον ε, μικρότερο τόνο σε ολόκληρο τον Ατλαντικό. Το 2009 εγκρίθηκε για να συμπεριληφθούν βασικά στοιχεία και μοντέλα αξιολόγησης επίσης, προκειμένου να συλλέγουμε επιστημονικά στοιχεία. Αυτό το πρόγραμμα είναι με 20 εκατομμύρια ευρώ, το 80% έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι για τέσσερα χρόνια. Για να τηρούμε την αρχή της διαφάνειας, η οποία διέπει, όπως είπαμε, όλες τις εργασίες της ΕΚΑΤ, όλες οι επιστημονικές εργασίες και όλη η διαχείριση που υπάρχει είναι στη διάθεση του κοινού. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στη συνέχεια τώρα, για λεπτά, Επίσης, ο κύριος Οντόναχιο, ειδικός από την Ένωση των Παραγωγών Αλλιευμάτων, Αλλιευτικών Προϊόντων, παλαιός φίλος της Επιτροπής Αλίας, ο κύριος Ντόναχιου. του δίνω το λόγο, λόγο για την παρέμβασή Thank you, uh, uh Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για ορισμένα πράγματα σε σχέση με τις οργανώσεις, περιφερειακές οργανώσεις αλίας. Φαντάζομαι ότι την ομάδα την οποία αντιπροσωπώ, που είναι η Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών, η προσοχή μας εστιάζει ε, στις περιφερειακές οργανώσεις αλίας η Λοιπόν, θα ήθελα ε, τα επόμενα λεπτά να σας εξηγήσω ορισμένα θέματα και ορισμένα είδη το οποίο αφοράν, αφορούν την Επιτροπή Ανατολικής, περιοχή Ανατολικής Περιοχής Αλίας και να σας πω τις δυσκολίες που έχουμε ως κλάδος με ορισμένα από αυτά τα προβλήματα και να καταλήξω σε συμπεράσματα, δηλαδή που πιστεύουμε ότι η ΝΙΑΦ μπορεί να λειτουργήσει. Θα έπρεπε ίσως να ρίξουμε μία ματιά στο χάρτη. Πού δραστηριοποιείται. Εδώ βλέπουμε στις ροζ περιοχές, τις τρεις διαφορετικές περιοχές της ΝΙΑΦ, ανατολικά του Ατλαντικού. Και από αλληλευτική άποψη δεν είναι αναγνωρισμένες αυτές τις περιοχές από τα ψάρια. Ε, ε, economic, ε, fishing zones. Και αυτό αποτελεί μέρος του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζουμε σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες. In terms of contracting parties, there are... Τώρα για τα συμβαλόμενα μέρη υπάρχει η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ρωσική Ομοσπονδία. Η Δανία ασχολείται με τις Φερόας νήσους και υπάρχει το Μπελίς, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία επίσης. Με δύο λόγια θα σας μιλήσω για το αντικείμενο της ΝΙΑΦ. Νομίζω ότι έχει σχέση με το ρόλο μας. Το αντικείμενο της ΝΙΑΦ είναι να συστήσει μέτρα για την ορθολογική αξιοποίηση του αλληλευτικού αποθέματος, λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Συμβούλιο για την ε, Διερεύνηση των Θαλασσών. Ως προς τα είδη που καλύπτονται από την ΙΑΦ, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο γάδος του Ατλαντικού, ο βακαλάος του Ατλαντικού, προσφυγάκι και όσον αφορά τα θέματα σε σχέση με την ΙΑΦ, η σύμβαση, σύμφωνα με τη σύμβαση, τα αποθέματά μας είναι καλά κατανεμημένα είναι ο Βακαλάος. Βλέπετε το χάρτη. Και τα, οι κίτρινες φυσαλίδες αλλιευμάτων που βρίσκονται γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Ορβηγία Από την Ορβηγία μέχρι την Ισπανία και μέχρι την Πορτογαλία. Συνεπώς τα αποθέματα είναι καλά κατανεμημένα. Ένας άλλος χάρτης που μας δείχνει τις μεταναστεύσεις, τις μετακινήσεις, το οποίο μας δείχνει ότι είναι καλά κατανεμημένα τα αποθέματα. Εδώ έχουμε τα προγράμματα διαχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιπροσωπεύει το 90% των αλλιευμάτων. We had agreed management arrangements between EU, Norway. Έχουμε ε, συμφωνία διαχείρισης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Νορβηγία Φερόες στη ζώνη που καλύπτεται από τη σύμβαση. Οι ροζ περιοχές που σας έδειξα. Αυτό ίσχυε μέχρι το 2009. Όλα όμω άλλαξαν από τότε που άρχισε να αναπτύσσει η Ισλανδία πολύ εκτεταμένη αλία και βλέπετε τους αριθμούς. Το 2001 δεν υπήρχε αλία στην Ισλανδία για τον Ατλαν... του Ατλαντικού. Το 2009 υπάρχουν αλλιεύματα πάνω από 130.000 τόνους. του 2006 τώρα. Ε, δεν έχουμε την τιμή μηδέν, αλλά το 2006 υπάρχει ένας ε, συντελεστής πολλαπλασιαστικός 31. Αν δείτε αυτούς τους αριθμούς, δεν είναι στοιχεία τα οποία παρουσιάζω εγώ, αλλά είναι ε, τα στοιχεία της ΙΖΕ. Θα δείτε εδώ ότι η Ισλανδία το 2006 είχε 1% και το 2009 22-24% ε, και αυτό είναι ε, τα αποθέματα πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλα. Συνεπώς, η βιωσιμότητα ενός αποθέματος απειλείται και πέραν αυτού υπάρχουν και οι Φερόες νήσοι. που αποσύρθηκαν από το μηχανισμό διαχείρισης του 2010 και προβλέπουν αλλιεύματα πάνω από 100.000 τόνους. Αλλά και η Ρωσία έχει μπει στο παιχνίδι σήμερα. έχουν ελευθερία αλίευση και συνεπώς θα μπουν μέσα στο παιχνίδι. Και προβλέπεται ότι θα αλλιεύσουν επιπλέον 40.000 τόνους ε, στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση, το οποίο σημαίνει περίπου 300.000 τόνοι πάνω από ε, το επιτρεπόμενο αλίευμα που συνιστάται. Αυτό είναι δυσβάστακτο. Πρέπει να αντιδράσουμε. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Ποιο θα αντιδράσει και πώ θα αντιδράσει. Δυστυχώ, η σύμβαση δεν έχει αρμοδιότητες, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να επιβάλλει κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία όμως μπορούν να δράσουν. Και προτείνω διάφορες λύσεις. Φυσικά θα θέλαμε να έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Βολευτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής. Υπάρχουν όμως μέτρα εμπορικής αλίας, ε, ε, το λόμπινγκ που γίνεται στο περιβάλλον, στις εξωτερικές υποθέσεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνουν τα πράγματα μόνα τους, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά τι συνέβη στο παρελθόν, όπου ο καθένας κάνει αυτό που θέλει στον τομέα της αλίας. Prior to 2006 we had we we had uh, uh, on constraint. στο προσφυγάκι υπήρχαν περιορισμένοι ε, υπήρχε περιορισμένη αλία. Τώρα πάλι αυτά τα αποθέματα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εάν δεν λυθούν τα προβλήματα ε, θα, θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Βλέπετε ότι και ε, η η αλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε ορισμένες ποινές, αλλά τώρα επειδή υπάρχει μείωση αποθέματος, ε, υπάρχει μείωση και δεν έχουν επιβληθεί ποινές. Υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν σχέση με την ΙΑΦ. Το Rockle Haddock. Για πολλά χρόνια προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα διαχειριστικό πρόγραμμα με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Διαπιστώνουμε όμως ότι τα αποθέματα του Καλαρία περιορίζονται εν μέρη επειδή δεν, η ρύθμιση αυτή δεν λειτουργεί. Επίσης, πρέπει να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κάνει η ΝΙΑΦ για τον έλεγχο αυτών των αλλιευμάτων. Κυρία Πρόεδρε, καταλήγω σε ορισμένα συμπεράσματα σε σχέση με την ΝΕΑΦΚΑ. Πιστεύουμε ότι δεν έχει εξουσίες η ΝΕΑΦΚΑ για να σταματήσει ε, την αδιάκριτη αλληλεία από τα μεμονωμένα συμβαλόμενα μέρη. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των παρακτήων χωρών. Αν λοιπόν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και επίσης υπάρχει το θέμα της ευθύνης των αλλιευμάτων. Είναι η ΝΕΑΦΚΑ που είναι υπεύθυνη ή οι χώρες. Αυτό το οποίο προτείνω είναι, όπως και με την κοινή αλληλευτική πολιτική, να αναθεωρήσουμε την ΕΑΦΚΑ, να δούμε ποια είναι η διακυβέρνησή της, να δούμε τις λειτουργίες της, τις εξουσίες της και τους σκοπούς της. Ευχαριστώ. Sí, muchísimas Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντόναχιο. στην συνέχεια ο τελευταίος που θα παρεύει είναι ο κύριος Γεωργάτε που θα αντικαταστήσει τον κύριο Μωρόν. Για λόγου ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί. Κύριε Γκαβάτε, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τα μέλη τη Επιτροπής ε, Αλίας και ανάπτυξη που όπω είπατε ο κύριο Μωρό δεν μπορούσε να προσέλθει αλλά μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω και με ιδιαίτερη χαρά. Στην εισήγησή μου θα αναπτύξω δύο κύριε ιδέε. Πρώτον, μια σαφή προάσπιση στον ε, τομέα τη αλίας, ε, των περιφερειακών οργανώσεων αλίας και από την άλλη πλευρά θα παρουσιάσω κάποιε προτάσει για το πώ μπορεί να βελτιωθεί ο σημαντικό αυτό ρόλο που έχουν οι περιφερειακέ οργανώσει Όπω σα έλεγα για τον τομέα, <clears throat> οργανώσεις αυτές ε, συμβουλευτικές ε, οργανώσεις αλίας είναι ο κύριος και σχεδόν μοναδικός μηχανισμός για τη διατήρηση και ε, διασφάλιση των μεταναστευτικών αυτών ειδών και αλλιευμάτων μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Ευτυχώς αυτό δεν είναι μόνο για τον αλλιευτικό τομέα έτσι που γίνεται, αλλά μπόρεσε να διαπιστωθεί και πρόσφατα στην διάσκεψη αναθεώρησης της Συμφωνίας της Νέας Υόρκης που έγινε πριν από μόλις ένα μήνα στη Νέα Υόρκη που ήμουν και παρόν εκεί σε αυτή τη διάσκεψη, μπορούσε να διαπιστωθεί ότι οι συστάσεις λοιπόν αυτής της διάσκεψης, σε αυτές αναφέρεται ο κύριος ρόλος των ΟΕΡΠ. Παρότι οι συγκεκριμένες οικολογικές οργανώσεις και ομάδες και κάποιες χώρες επέκριναν και έντονα και όλα στον ρόλο αυτών των περιφερειακών οργανώσεων αλλίας, παρόλα αυτά στις συστάσεις, γιατί υπήρχε ευρύτατη πλειοψηφία, αντανακλώταν αυτό και είχε συμπεριληφθεί όταν ε, συνέβη αυτή η ε, συνεδρία. Είναι πολύ εύκολο σκέφτηκα να ασκεί κανείς επικρίσεις όταν δεν έχει κανείς ε, στόλο, αλληλείας ή ζώνες που να αφορώνται άμεσα από τέτοιες επικρίσεις. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι παρόδο στο περιθώριο. Κατέστη σαφέ ότι για μα ε, οι περιφερειακέ οργανώσει αλληλεία έχουν κύριο ρόλο. Πρέπει επίση να δούμε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει αυτέ τι δραστηριότητε. Και αφενό έχουμε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο τη Θάλασσα και αφετέρου έχουμε τη Συμφωνία τη Νέα Υόρκη. Τη Συμφωνία τη Νέα Υόρκη για τα άκρο μεταναστευτικά είδη που είναι το Fish Stocks Agreement στα αγγλικά με τα αρχικά αυτά είναι γνωστό. Και έχουμε και δεοντολογικό κώδικα της ε, ΦΑΟ και ε, της ε, συναφής ρυθμίσης. Όλα αυτά τα αναφέρω επειδή δεν το γνωρίζουν όλοι και δεν έχουν εξοικειωθεί. Και όταν λέω σε όλους αναφέρομαι σε σχέση με αυτή την σύμβαση και που στον αλλιευτικό κόσμο εμείς ζητάμε από όλες τις χώρες να κυρώσουν και να ε, εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις. Ως επιχειρηματίες αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σταθερό πλαίσιο. Ένα αξιόπιστο σταθερό πλαίσιο που θα δίνει νομική ασφάλεια και να έχουμε σαφείς κανόνες που δεν θα αλλάζουν διαρκώς. Σε αυτούς τους σαφείς κανόνες συμφωνούμε να είναι σχέδια διαχείρισης ή ανάκαμψης μακροπρόθεσμα των αλλιευμάτων μέσω αυτών των περιφερειακών οργανώσεων αλλίας. Εν τέλει, εν κατακλείδη, αυτές ε, οι διατάξεις να εφαρμόζονται εξίσου σε όλα τα μέλη, σε όλα τα συμβαλόμενα μέρη, τους ε, εμπλεκόμενους και ή δυνατόν σε όλους εκείνους που δεν είναι μέλη για διάφορους λόγους. Εν τέλει, αυτό που χρειαζόμαστε είναι, όπως λέγεται στα αγγλικά, a level playing field, δηλαδή ένα δίκαιο ε, παιχνίδι, ένα συνθήκες ανταγωνισμού θεμητές. Θα ήθελα τούτου λεχθέντος να αναφέρω με σαφήνεια το εξής. Αν όλοι συμφωνούμε βέβαια ότι οι περιφερειακές οργανώσει αλληλεία είναι οι πιο σημαντικοί μηχανισμοί, εκείνο που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε είναι να αναζητηθούν προβλήματα ώστε να υπάρξουν, να προσκόμματα για τις διαφορετικές αλληλείε, διαφορετικές μορφές αλληλεία. Και όταν λέω τέτοιου είδου προσκόμματα ή εμπόδια, Έχω υπόψη κάτι το οποίο συνέβη εφέτες, εφέτος για τον ερυθρόπτερο τόνο και τις ΣΥΤΕΣ. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που έκανε το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, δεν, σε σχέση με τον αλλιευτικό τομέα, με τους αλλιείς, ήταν προβληματικό διότι διακυβεύθηκε η ύπαρξη και η συνέχεια της ΙΚΑΤ, που είναι μια οργάνωση η οποία για το καλύτερο ή το χειρότερο μπορεί να εργαστεί, μπορεί σίγουρα να βελτιωθεί. Μπορεί να βελτιωθεί αν τα κράτη που είναι τα μέλη της ε, ΚΑΤ και που είχαν τοποθετηθεί υπέρ της ε, ΣΥΤ σεβαστούν τις διατάξεις και κάνουν προσπάθειες να υλοποιηθούν οι διατάξεις. Γιατί όλα τα άλλα θα είναι δημαγωγικά και θα είναι δημαγωγία που δεν θα εξυπηρετεί τίποτα. Έτσι λοιπόν το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε σχέση με τον τομέα και την Ευρωβουλή είναι να μην δημιουργηθούν προβλήματα και να ε, στοιχηματίσετε υπέρ των περιφερειακών οργανώσεων αλληλεία και στα πραγματικά πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ευτυχώ οι περιφερειακέ οργανώσει αλληλεία πρόοδευσαν και βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό στον τρόπο δράση του και στον τόπο, τρόπο διοργάνωση των εργασιών του τα τελευταία χρόνια. Και αυτό αναγνωρίστηκε και από τα Ηνωμένα Έθνη πρόσφατα. Και πέρα από τι ε, κριτικέ και επικρίσει, επίση υπήρξαν πολλοί έπαινοι γιατί βελτιώθηκαν πολλά πράγματα. Βελτιώθηκαν οι διατάξει εσωτερική λειτουργία Πολλές ε, τέτοιες ε, περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας έχουν ε, αναδιοργανωθεί εσωτερικά, είναι τώρα πολύ πιο διαφανείς από ό,τι στο παρελθόν Επίση, ε, ασχολήθηκαν με την προστασία των ευάλωτων οικοσυστημάτων. Αναζητήθηκαν σοβαρά μέτρα προστασία ε, του περιβάλλοντο. και σε σχέση με τι ε, οργανώσει για τον τόνο και μέσα στη διαδικασία κόμπε, όπω είναι γνωστή, υπάρχει συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών περιφερειακών οργανώσεων αλληλεία για να υπάρξουν συμφωνίε συντονισμού και εναρμονισμού. Και όλα αυτά αντανακλώνται, όπω ανέφερα, στην αναθεώρηση τη συμφωνία Νέα Υόρκη, που πριν μόλι από ένα μήνα διεξήχθη στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, Παρόλα αυτά, αφενό, πολλά μπορούν να γίνουν για να βελτιωθούν τα πράγματα και δεν πρέπει να δημιουργηθούν προβλήματα και προσκόμματα. Χρειαζόμαστε τη δέσμευση και εμπλοκή όλων για να ενισχυθούν αυτέ οι περιφερειακέ οργανώσει Πώς Πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρώτον. Με, κράτη τα οποία θα δεσμεύονται περισσότερο και θα είναι πρωτοπόροι και θα έχουν πολιτική βούληση, όχι μόνο να υιοθετούν τις διατάξεις που θα προτείνονται σε σχέση με τις περιφερειακές οργανώσεις ε, αλληλείας, αλλά θα τις υλοποιούν και θα τις υλοποιούν με σοβαρό πνεύμα και τρόπο. Δεύτερον, πρικοδοτώντας τις γραμματείες αυτών των οργανώσεων με περισσότερα στελέχη, περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό και κονδύλια, αλλά και επιστημονικά, επιστημονική υποστήριξη και ενίσχυση. Είναι ένα από τα ε, προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτέ οι περιφερειακές οργανώσει αλλιέ, Θα επανέλθω στη συνέχεια σε αυτό το θέμα. Επίση, και αναφέρθηκε προηγούμενα, χρειαζόμαστε ένα σύστημα ελέγχου, το οποίο θα είναι πολύ πιο διαφανέ, πολύ πιο σαφέ και ε, ευδιάκριτο και με την ανάγκη να χρησιμοποιούνται, να εφαρμόζονται κυρώσει σε εκείνους που δεν θα τηρούν τα υπεσχημένα. Αν κάτι έχει ε, συμφωνηθεί, σε σχέση με την ε, υλοποίηση και συμμόρφωση, αν δεν υπάρχουν ε, κάποια μέτρα και δεν υπάρχουν κυρώσεις, τότε δεν θα ε, υπάρχει κανένας λόγος ύπαρξη αυτών των διατάξεων. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συλλογή δεδομένων και στοιχείων και επιστημονικών στοιχείων σχεδόν σε όλες τις οργανώσεις, περιφερειακές οργανώσεις αλίας. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα όπω η ΝΑΦΟ και ε, επίσης μετά από χρόνια ε, προσπαθειών για την ανάκαμψη των αλλιευμάτων έγιναν τεράστιες προσπάθειες να μειωθεί η αλλιευτική προσπάθεια και να αφαιρεθούν σκάφη, να μειωθεί ο στόλος και καταδείχθηκε σε σχέση με την, ε, το πρότυπο αυτό δεν ήταν το πιο κατάλληλο στο παρελθόν και είχαμε στοιχεία εσφαλμένα και λανθασμένα. Τώρα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που συναποτελούν μέρος αυτών των περιφερειακών οργανώσεων αλλιεύσεων πρέπει να επενδύσουν έχει αναφερθεί αυτό πολλέ φορέ και στο Ευρωκοινοβούλιο και σε άλλα φόρα. Πρέπει να επενδύσουν σε δράσει έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα. Αν δεν το κάνουν αυτό, οι διαχειριστέ θα πρέπει να λάβουν αποφάσει χωρί να έχουν επαρκή τεκμήρια και επιστημονικά στοιχεία και πιθανόν θα λάβουν λάθο αποφάσει. Όπω έγινε πιο πριν, για παράδειγμα, με το ε, προηγούμενο αλίευμα που ανέφερα. Και έτσι πρέπει να ενισχύσουμε τη σημαντική παρουσία των Ευρωπαίων επιστημόνων στα διάφορε επιστημονικέ επιτροπέ. Δεν είναι δυνατόν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντα συνειδητοποιήσει βέβαια τα όρια που υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να προσέρχονται οι επιστήμονε σε αυτή την Επιστημονική Επιτροπή λόγω έλλειψη κονδυλίων. Κάτι τέτοιο δεν είναι λογικό και συνετό και τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να το συνειδητοποιήσουν αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά τη πρέπει να υποστηρίξει αυτά τα κράτη-μέλη για να μπορούν να αποστέλουν αυτού του επιστήμονε το επιστημονικό προσωπικό και σίγουρα αυτό θα συνεισφέρει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Απ' την άλλη πλευρά είναι ανάγκη να ενιοποιηθούν, να εναρμονιστούν υποχρεώσει υποχρεώσεις από τα διάφορα συμβαλώμενα μέρη. Ιδιαίτερα θα θέλαμε εμεί να γενικευθούν τα μέτρα τα οποία ήδη υφίστανται σε σχέση με τον κοινοτικό στόλο να επιβληθούν στου άλλου στόλου που ανταγωνίζονται με εμά στα ίδια ύδατα και τα οποία ε, υπορρύθμιση αυτών των οργανώσεων αλληλεία θα πρέπει να βρίσκονται γιατί αφορετικά θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα θέμη του ανταγωνισμού σε σχέση με του υπόλοιπου ε, που ανταγωνίζονται την, ε, στόλου τη της Ένωσης. Μια άλλη πτυχή που μπορεί να βελτιωθεί και είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνει σε όλε τι περιφερειακέ οργανώσει αλληλεία η επαρκή διαχείριση του δυναμικού του στόλου. Δεν θα επισέλθω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να παγωθούν, αν θα πρέπει να παγωθούν να αυξηθούν ή να μειωθούν. Εκείνο που πρέπει να γίνεται είναι σε σχέση με ε, το δυναμικό κάθε στόλου και τα αλλιεύματά του να εξευρεθεί αναγκαία ισορροπία. Σε κάποιε περιπτώσει ε, δεν συμβαίνει αυτό βέβαια. Και μέλη, αξιότιμα μέλη αυτής της Συγνωβευτικής Επιτροπής αλληλία και ανάπτυξη. Ε, δεν πρέπει να ντρέπεται κανείς ή να φοβάται να προασπίζει τα συμφέροντα του κοινοτικού ε, στόλου και των κοινοτικών αλλιέων σε αυτές τις περιφερειακές οργανώσεις αλλιέας. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα θεμητά συμφέροντα του τομέα έναντι προτάσεων που καμιά φορά δεν έχουν ούτε και τεχνική δικαιολογία, ούτε και επιστημονικά βάθρα. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να υπερασπιζόμαστε εκείνες τις επιχειρήσεις και Ευρωπαίους εργαζόμενους που ασχολούνται με την αλληλεία. Και πρέπει να το γνωρίζουμε και το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό, γιατί καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι κάποιοι έχουν ντρέπονται να υποστηρίζουν ή να υπερασπίζονται τον αλληλευτικό τομέα του αλληλεί λόγω των πιέσεων που υφίστανται. Για την βελτίωση επίση τη λειτουργία των περιφερειακών οργανώσεων αλληλεία πρέπει να διατηρηθεί ένα σύστημα άμεση διαβούλευση με τον αλληλευτικό τομέα Αποστέλλοντα τι προτάσει στον τομέα μέσα σε έγκαιρες προθεσμίες, με επαρκή χρονικό, επαρκές χρονικό διάστημα για να μπορούμε να τα μελετήσουμε, να τα ε, μελετήσουν και οι εφοπλιστές και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν τα πράγματα. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των δυνατοτήτων βελτίωσης που μπορούν να γίνουν και μέσα από τη διαδικασία του ΚΟΜΕ, πρέπει να συσφιχθούν οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών περιφερειακών οργανώσεων αλλία, όχι μόνο για τον τόνο, αλλά και για, τις άλλες, για τα άλλα είδη δημιουργώντα εγκάρσια οριζόντια θέματα με εναρμονισμένα μέτρα που σίγουρα θα διευκολύνουν τη λειτουργία και τη δράση των εμπλεκόμενων. Για αυτού του λόγου, έχοντα τοποθετηθεί και έχοντα πει ποιε είναι οι βελτιώσει που εμεί θεωρούμε ότι μπορούν να εισαχθούν, Μία πτυχή που πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει σαφώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Είναι ένα ρόλο προπομπού, πρωτοπόρου, όπου φυσικά πρέπει να διασφαλιστεί η αηφορία στην αλληλεία και η βιωσιμότητά της και να δρώσουμε με, με συνεκτικότητα και συνέχεια. Και δεν είναι δυνατόν από μια... τη μια πλευρά να <laughs> προσπιζόμαστε τις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας και μετά να αντιστρέφουμε τα πράγματα και να ε, αντιβαίνουμε τα όσα έχουμε συμφωνήσει με άλλες δράσεις και γι' αυτό θα πρέπει να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις ε, όσον αφορά την κατεύθυνση που ε, υπερασπίζονται οι περιφερειακές οργανώσεις αλλίας και αν θυμάμαι καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Ιαπωνία είμαστε εκείνοι που είμαστε παρόντες στις περιφερειακές οργανώσεις αλλίας σε όλες αυτές και είμαστε λοιπόν ένα σημείο αναφοράς παγκόσμια. Και χωρί αμφιβολία, αυτά τα οποία θέλω να πω με αυτά είναι ότι η πολιτική επιρροή τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνάδει και να είναι παραλίλου να βαίνει με την οικονομική επιρροή και δύναμη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προωθήσουμε, να προαγάγουμε τι σχέσει μα με τρίτε χώρε, ιδιαίτερα με εκείνε για τι οποίε υπάρχουν συμφωνίε σύνδεση και για την αλία, για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τι αλληλευτικέ προσπάθειε στι περιφερειακέ οργανώσει αλία. Ολοκληρώνω, Πρόεδρε. Υπογραμμίζοντα την σημασία που για μα έχει το να βασιζόμαστε σε ένα ευρωπαϊκό στόλο <clears throat> ε, εκτός υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα, είναι, μπορεί να συναγωνιστεί και σε, διαφορά, σε ε, αντίστοιξη με την Πράσινη Βίβλο και σε σχέση με τα, ε, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την οδό που είχαν ακολουθήσει σήμερα τουλάχιστον θεωρείται σημαντικό να υπάρχει αυτός ο κοινότικό στόλος. Διότι έχουμε αυτή τη διαφορά, όπως είπε ο Άλμπερτ Άινστάιν, και αυτό το είπε και ο Μωρόν πριν από πέντε χρόνια, το να δίνει κανείς ε, το παράδειγμα δεν είναι μόνο ο κύριος τρόπος να επηρεάζει τους υπόλοιπους, είναι ο μόνος τρόπος να είναι κανείς το καλό παράδειγμα. Και αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Στόλος ε, για τους υπόλοιπους. Και εν τέλει, για να ολοκληρώσω αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να πω ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ενότητα, η ένωση των ε, περιφερειακών οργανώσεων αλληλείας. Διότι βρισκόμαστε σε όλες τις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας, είμαστε πολύ ε, είναι πολύ λίγοι οι υπάλληλοι και δεν μπορούν να πηγαίνουν παντού παγκόσμια και είναι δύσκολο να μπορεί κανείς να, καλύψει το έργο που έχει να επιτελέσει με λίγα στελέχη, με λίγους υπαλλήλου. Πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν το συντονισμό όπως προαναφέρθηκε σε σχέση με την ανάπτυξη, το εμπόριο, την υγεία, την υγειονομική πολιτική και την πολιτική για το περιβάλλον φυσικά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Παρακαλώ τώρα. Ξεκινάει η συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές μας για τις απόψεις που εξέφρασαν και θα ξεκινήσω από το τέλος, θα ξεκινήσω από την τελευταία παρουσίαση. Πιστεύω ότι εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε δείξει ότι στηρίζουμε τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας. Αυτό φαίνεται από το κείμενο τη κοινή ελευθερική πολιτική, παρόλο που πρέπει φυσικά να εντατικοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τι προσπάθειέ μα για τα επόμενα κείμενα. Δύο θέματα. Το επιστημονικό κριτήριο. Τα κοινά κριτήρια, οι κοινέ αξιολογήσει και από την άλλη μεριά πιστεύω ότι χρειάζονται και από την άλλη μεριά στηρίζουμε τι περιφερειακέ οργανώσει αλλία να κάνουν προτάσεις λογικές, αξιόπιστες, με συνένεση, με διαφάνεια, όπως υπόθηκε εδώ. Στηρίζουμε λοιπόν τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας γιατί μπορούν να προσφέρουν επιτόπου λύσεις. Δεν στηρίζουμε την αποκέντρωση της ε, κοινή ελευτικής πολιτικής. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό από εδώ. Η αυτάρκεια είναι θέμα που πρέπει πιο συγκεκριμένα να εξεταστεί σε μια πιο ειδική συζήτηση, πιστεύω. Θέλω επίσης να ρωτήσω κάτι την κυρία Παγιαρές, η οποία μας εξήγησε τη λειτουργία της ΙΚΑ. Επίσης, μας εξήγησε ποιες είναι οι δράσεις για τα τονοειδή. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση, λοιπόν. Όταν μιλάμε για το μακρύτερο τόνο και μιλάμε για την παράνομη ελεία. Πιστεύετε ότι με τα μέτρα τα οποία εσείς θέτετε για τον έλεγχο, για τα ειδικά προγράμματα, για τους παρατηρητές, για έλεγχο των εκφορτώσεων, για τον έλεγχο με παρατηρητές επιτόπου εκεί που γίνεται η πάχυνση των ηχθείων, πιστεύετε ότι μπορεί να ελεγχθεί η παράνομη αλία στα λιμάνια ή στα σκάφη που είναι πάνω από 24 μέτρα. Πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί αυτό. Τι πιστεύει η ΚΑΤ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λουβίν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όσους μίλησαν. Θα συνεχίσω στα αγγλικά, επειδή θα διαβάσω μια έκθεση της ΙΚΑΤ όσοι γνωρίζουν την ε, ΕΚΑΤ, Νομίζω ότι είναι μια έκθεση του 2008 και μας λέει ότι η αξιολόγηση της απόδοσης ε, της ΕΚΑΤ για τη διαχείριση της αλίας ε, του τόνου, κυρίως στον Ανατολικό Ατλαντικό και στην Μεσόγειο, θεωρείται ως μια ντροπή διεθνώς και η διεθνής κοινότητα η οποία ανέθεσε τη διαχείριση αυτών των εικονικών ειδών στην ΑΕΚΑΤ θα έπρεπε ε, να, ε, να έχει φροντίσει η ΑΕΚΑΤ να χειριστεί καλύτερα το θέμα. Αυτό είναι σκληρό. Η αξιολόγηση όμως κατονομάζει κυρίως τις ε, τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή τις χώρες που συνεργάζονται στα πλαίσια της ΕΚΑΤ και όχι στη γραμματεία της ΕΚΑΤ. Θα ήθελα όμως να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της ΑΕΚΑΤ. Τι μέτρα έχουν ληφθεί από τότε που έγινε αυτή η αξιολόγηση ώστε να βελτιωθεί η απόδοση η επίδοση της ICAT. και κυρίως εκείνη ε, των ε, συμβαλωμένων χωρών. Δεν αρκεί να έχουμε κείμενα. Πρέπει να υπάρχει και συμμόρφωση στα κείμενα. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Και έρχομαι τώρα στο επόμενο ερώτημα. Πιστεύετε ότι η ICAT έπρεπε να προβλέπει περισσότερες κυρώσεις, ώστε να φροντίζει οι χώρες να συμμορφώνονται με τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Και το ερώτημά μου είναι κατά πόσον αρκεί η ΆΙΚΑΤ για να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες. Ο κ. Γκαράτ επίσης αναφέρθηκε σε όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η διεθνής κοινότητα και επίσης ε, το ε, δίκαιο της θαλάσσης ε, του ΟΗΕ και επίσης οι ελευτικές συμφωνίες. Όλες αυτές οι συμφωνίες είναι θαυμάσιες στα χαρτιά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι περισσότερες χώρες δεν εφαρμόζουν τις συνθήκες. Γι' αυτό παρακαλώ να μου πει ο κ. Γκαράτ και επίσης και ο εκπρόσωπος της ICAT αν πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ανώτερο όργανο σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών το οποίο καταρχήν θα αξιολογεί την επίδοση των FMOs και δεύτερον, εάν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το Διεθνές Δικαστήριο του Δικαίου της Θαλάσσης, ώστε να εφαρμοσ... να τηρούνται οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτές τις συμφωνίες και τελικά να λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά όταν πρόκειται ε, για τις διεθνείς συμφωνίες, για τα μεταναστεύοντα αλλιευτικά αποθέματα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό στο διεθνές σύστημα ε, ως προς την παρακολούθηση και την τήρηση των συμφωνιών. Άλλωστε είδαμε τα αποτελέσματα και με τον τόνο. Εδώ έρχομαι σε ένα άλλο ερώτημα ε, για τον εκπρόσωπο της ICAT. Επειδή πάντοτε μιλάμε για τον τόνο, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη τα οποία προβλέπονται και τη διαχείρισή τους έχει αναλάβει ΆΙΚΑ, ο τροπικός τόνος και είδαμε και το πρόβλημα. Ε, είδαμε τις κουκίδες, τις κόκκινες κουκίδες στην παρουσίασή σας. Υπάρχουν και πολλά είδη, άλλα είδη, των οποίων η διαχείριση δεν είναι ευτυχή. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά. Και τέταρτον, θα ήθελα να μιλήσω για την κατανομή των αλλιευτικών πόρων. θεμητά αιτήματα υπάρχουν από τι αναπτυσσόμενες χώρες που λένε ότι δεν υπάρχουν ιστορικά αλλιεύματα για ορισμένα μεταναστεύοντα αλλιευτικά αποθέματα. Αλλά τώρα με την ανάπτυξή τους θέτουν το ερώτημα και ζητούν να τους δοθεί μέρος αυτών των αλλιευμάτων που, που μπορούν να αλλιεύονται. Και παρακαλώ τον κύριο Γκαράτ να μας πει τη γνώμη του τι πιστεύει για αυτά τα αιτήματα και τι πρέπει να κάνουμε σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, ο κ. Γκαράτ, ως εκπρόσωπος της, της Ένωσης που μας παρουσίασε, νομίζετε ότι ε, οι φορείς που υποδείχθηκε ότι αλλιεύουν νόμιμα μπορούν να έχουν το δικαίωμα να αλλιεύουν στα πλαίσια των RFMOs. Και τέλος, στρέφομαι στον κύριο Ντόναϊου, ο οποίος μα μίλησε για την υπεραλία για το προσφυγάκι. Σε ποιες χώρες έγινε αυτή η αλία στο προσφυγάκι, η υπεραλία. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Ο Γκάλαγκερ. Ευχαριστώ. Άκουσα τους ομιλητές και κυρίως τον κύριο Οντόναχιου από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Ενώσεων Παραγωγών Αλίας. Εκείνος λοιπόν μας είπε αυτά που μας είπε και ο Νορβηγός σήμερα το πρωί και ο κύριος Πάσαρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ότι δηλαδή με τα χρόνια προσπαθούμε να έχουμε μια βιώσιμη αλία, αλλά το προσφυγάκι ή το σκουμπρί. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ό,τι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις έχουμε. Οι χώρες προσπαθούν πια ε, να λειτουργήσουν μαζί γιατί αλλιώς θα κλείσει η αλία. Και τότε αρχίζει και ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα όμως το έχουμε. Το κουδούνι του συναγερμού έχει χτυπήσει. Πρέπει να το ακούσουμε. Ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην είναι σε ισχυρή θέση για να κάνει ό,τι πρέπει να γίνει, αλλά μην τι άλλο να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και αυτούς που μας εκπροσωπούν να αναλάβουν ό,τι δράση χρειάζεται. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για την αλία. Και άλλε δράσεις μπορούν να ληφθούν. Σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ ώστε και άλλες χώρες, οι παράκτιες χώρες, να δρουν και αυτές υπεύθυνα. Ακούστηκε η διακυβέρνηση, οι εξουσίες, όλα αυτά πρέπει να τα φροντίσουμε και όχι σε ένα χρόνο, τώρα. Αυτό δηλαδή που μας λέω, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι δεν μπορεί να καθόμαστε εδώ και να ακούμε, με κάθε σεβασμό σε όσους πήραν το λόγο, τους ακούμε και μετά θα ξανάρθω και θα του ξανακούσουμε. Εγώ ελπίζω πριν το καλοκαίρι, τέλος πάντων πριν από την επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε, να βρεθούμε στο κυκλισμένο το θυρών μεταξύ μα και να πούμε τι δράση πρέπει να αναλυφθεί προκειμένου να έχουμε μία αλία. Γιατί εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την ε, αλία, φυσικά, αλλά αυτό να γίνεται με βιώσιμο τρόπο. δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις, γιατί αλλιώς το μέλλον θα είναι σκοτεινό. Το μέλλον τώρα είναι στα χέρια μας, όχι μόνο στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα χέρια ολωνών. Να πάρουμε λοιπόν ό,τι μέτρα πρέπει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, αλλά ειλικρινά αυτή τη δήλωση ήθελα να την έχω κάνει. Και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Κάλεγερα. Η κυρία Ρομπούστο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Πρέπει όμως ιδιαίτερα να πω ότι σε σχέση με το τελική παρατήρηση του κυρίου Γκάλακερ θα μπορούσε κανείς το συμπέρασμα να το πάρει αυτό. Αυτό πρέπει να κάνουμε, θα μπορούσε κανείς να πει. Το θέμα είναι πότε, πώς και πόσο γοργά. Έχουμε το πρόβλημα ότι έχουμε διαφορετικές τοποθετήσεις για επιχειρήματα. Γι' αυτό ερωτώ τους, τον εκπρόσωπο των Περιφερειακών Οργανώσεων Αλληλείας πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα των σημεών ευκαιρίας Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τις σημαίες ευκαιρίας ε, όσον αφορά του στους αλληλευτικούς στόλους. Και στον άλλο εκπρόσωπο θα ήθελα να πω ότι έχω διαβάσει ένα δημοσίευμα στον τύπο ότι επικρίνεστε από την Greenpeace ότι οι ίδιοι εσείς στον Δυτικό Ειρηνικό είχατε αλλιεύσει λέει παράνομα. Μπορείτε να μας πείτε κάτι ακριβέστερο για αυτό το στοιχείο. Είναι μια, μια επινόηση της ε, Greenpeace, ένα μύθευμα το οποίο έχει καθ' υπερβολή ε, διονγκωθεί. Υπάρχει κάτι πίσω από όλη αυτή την ιστορία, μήπως ε, κάποια δίκη ή κάποια νομική διαδικασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος να παρέμβει αυτή τη στιγμή. Θα κάνω κι εγώ ένα σχόλιο επίσης. Προσέξτε, οι περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας ε, προφανώς δεν είναι οργανισμοί που να λειτουργούν με τέλειο τρόπο και όλοι εδώ έχουν κάνει και επικρίσεις ε, όχι μόνο σε σχέση με τις ε, ε, δράσεις αυτές αλλά σίγουρα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο ξεκινώντας να αναδιοργανώσουν τις εμπορικές αυτές πτυχές που αφορούν την αλία στα κοινοτικά ύδατα και στα διεθνή ύδατα. Και ένα θετικό στοιχείο που, διοργανώ, που τις χαρακτηρίζει είναι και όλας και η πολυπλοκότητα και ο μεγάλος αριθμός των συμβαλωμένων ε, μερών. Έχουμε αναπτυσσόμενα κράτη που έχουν δυσκολίες ε, για να υλοποιήσουν τα μέτρα και τα λοιπά και να συμμορφωθούν έτσι σε κάποιες διαδικασίες υπάρχουν βραδύτεροι ρυθμοί από ό,τι επιθυμούσαμε και αυτό επίσης αληθεύει. Όμως είναι πρόδειλο ότι αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι τα Ηνωμένα Έθνη σε πολλές ε, άλλες ε, διασκέψεις και συνόδους έχουν ε, εντοπίσει και έχουν εκφράσει την, το ενδιαφέρον τους και υποστηρίζουν τις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας όσον αφορά βάλλοντα είδη κτλ. Λοιπόν, είναι θα έλεγα το το έλασον από πλευράς αρνητικών στοιχείων για την ε, προώθηση των συμφερόντων των ε, ε, αλλιευτικών τομέων. Επίσης, για τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας, που είναι οι οργανισμοί όπου βρίσκονται οι διαχειριστές ε, των ε, ειδών αυτών, κάθε ένας ε, για λογαριασμό του και υπάρχουν και οι επιστήμονες, επιστημονικοί ερευνητές, παρότι δεν είναι πλήρης αυτή η επιστημονική έρευνα. Και σε αυτοί θα είναι οι τελευταίοι που θα πρέπει να λάβουν τις τελευταίες συστάσεις ή τις τελευταίες αποφάσεις ή και σε σχέση και με άλλους οργανισμούς, τα κτλ. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να γίνεται είναι να λέγεται ότι η ΚΑΤ, η ΝΕΑΦ, η ΕΝΑΦΗ ή οποιοδήποτε άλλο είναι οργανισμό που θα διαχειριστεί αλλιευτικού πόρου και μετά όταν κάποιος, σε κάποιον δεν αρέσει κάτι να πούνε Α, θα πάμε σε άλλον. Εμεί θα πάμε στη σύνθεση σε κάποιον άλλο. Είναι ένα πρόβλημα. Πέρα από το ότι τίθεται πρόβλημα για το μέλλον και για το πώ θα διαμορφωθούν αυτά τα πράγματα, σε ποια πλαίσια και σε σχέση με τις ε, επισημάνσεις από πλευράς ε, ε, άλλων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας ε, είναι οι οργανώσεις που θα πρέπει να επιλαμβάνονται αυτών των θεμάτων. Μετά πάνε τα θέματα αυτά και προστρέχουν στις ΣΥΤΕΣ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι σε σχέση με αυτό και για τις ΣΥΤΕΣ και για τον ερυθρόπτερο τόνο δεν είναι μια οργάνωση που προβλέπεται για εμπορικά είδη Μάλιστα υπάρχει και έλλειμμα ερευνητικό και γι' αυτό ζητεί από την ΦΑΟ και υπάρχει σύμβαση σε σχέση με τη ΦΑΟ ώστε μια επιστημονική επιτροπή να υποστηρίζει και να συνδράμει Α, όχι, εντάξει. Έχει μια συμφωνία με τη ΦΑΟ, ώστε μια επιτροπή επαϊόντων αξιωματούχων να τους συνδράμει για να δουν αν θα, είναι, θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα παράτημα ή όχι αυτά τα είδη. Γι' αυτό αυτό που λέω είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι καλύτερα προετοιμασμένες οι, οι ε, οργανώσεις, περιφερειακές οργανώσεις αλίας σε σχέση για παράδειγμα με άλλα είδη από ό,τι για τον ερυθρό τόνο. Αυτό θα ήθελα να θέσω σε ερώτημα και περνάμε στις άλλες παρεμβάσεις και με τη σειρά θα πάρω τον λόγο η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΑ που εκπροσωπείται εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του κυρίου Δήμου για να μπορέσει να ολοκληρώσει με τις ε, παρεμβάσεις τα στοιχεία αυτά που έχουμε. Η κυρία Παγιάρέ όμως θα λάβει πρώτα τον λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα απαντήσω από κοινού στην πρώτη κατηγορία, πρώτη ομάδα αυτών των ερωτήσεων που επικεντρώνονται στον ερυθρόπτερο τόνο ουσιαστικά. Ο ερυθρόπτερος τόνος μετά την αξιολόγηση του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνήθεται το 2009 υιοθέτησε μια σύσταση που ανέφερε, ε, μείωνε σε 50% το μέγιστη, μέγιστη αλίευση κατόγκων και έλαβε σημαντικά μέτρα ελέγχου μεταξύ αυτών όπως και προανέφερα στην παρουσίασή μου το Περιφερειακό Πρόγραμμα Παρατηρητών για τον Ερυθρόπτερο Τόνο που σημαίνει ότι όλες οι ε, δράσεις ε, σε σχέση με την αλία θα ε, υπεβάλλοντο όσον αφορά τις, ε, τον γρήπο ή και τις ε, μονάδες πάχυνσης που είναι τα δύο θα έλεγα επίκεντρα με τη μεγαλύτερη επίπτωση όσον αφορά αυτού του είδους τα λιεύματα θα βρισκόντουσαν πάντα, θα είχαν πάντα την παρουσία εποπτών. Και για αυτό το έτος υπήρχε μια πολύ συντομότερη περίοδος από ό,τι είχε προβλεφθεί, διότι λόγω των συστημάτων εποπτείας διαπιστώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν ε, οι ποσοστώσεις και μετά σταμάτησε η αλληλευτική προσπάθεια. Το ίδιο συνέβη και σε σχέση με τους γρίπους ε, όπου έχοντας ξεπεράσει τώρα ε, αυτές τις ποσοστώσεις απελευθερώθηκαν από αυτή τη δραστηριότητα. Και παρομοίως σε σχέση με, με την εποπτεία για τις, ε, την παράνομη αλληλεία επίσης, την εποπτεία σε σχέση με τις ε, ε, παράνομες αλληλευτικές δράσεις και σε σχέση με το 98% των αλλιευμάτων που προέρχονται από συμβαλόμενα μέρη ή συνεργαζόμενα μέτρα, μέρη, η ε, αναλογία θα έλεγα είναι σε σχέση με άλλες περιφερειακές οργανώσεις πολύ μικρή που βασίζονται σε πολύ μικρότερη συμμετοχή συμμετεχόντων και συμβαλωμένων μερών όσον αφορά τους ε, αλληλείς. Σε σχέση με... Και πάλι τώρα εδώ όσον αφορά τον ερυθρόπτερο τόνο. Την προηγούμενη Κυριακή κιόλα ε, ολοκληρώθηκε μια προπαρασκευαστική συνεδρίαση όσον αφορά τα στοιχεία των ερυθρόπτερων τόνων για την μελλοντική αξιολόγηση που θα γίνει το Σεπτέμβριο για τα αποθέματα και, στο και στη Δυτική και στην Ανατολική Μεσόγειο και όπως πάντα ήταν συνεδριάσεις ε, απόλυτα ανοιχτές, ανοιχτού χαρακτήρα για συμμετοχή από παρατηρητές και όπως και η συνεδρίαση για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, όλες οι αναλύσεις, όλες οι εκθέσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα και είναι προσπελάσιμες ε, για οποιονδήποτε επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία όσον αφορά την αναθεώρηση για την ε, περαιτέρω εξέλιξη των πραγμάτων για την ε, ΑΕΚΑΤ, τρει ανεξάρτητοι επαείοντε ε, και που δεν υπήρχε κάποια δέσμευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αποτελέσματα έχουν συμπεριληφθεί στις μελέτες και αυτή την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει μια συνάντηση για τον Λευκό Τόνο στη Μεσόγειο που ήταν ένα από τα σημεία τα οποία χαρακτήρισαν την αναθεώρηση σε αυτή την προσπάθεια. Ένα απόθεμα που λόγω έλλειψης, απουσίας στοιχείων δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης από την ΑΙΚΑΤ. Και για τις υπόλοιπες ομάδες όπως προαναφέρθηκε, η ομάδα για το μέλλον της ΙΚΑΤ που τέλη Ιουλίου θα συνέρθει στη Βραζιλία και που θα εξετάσει θέματα που συσχετίζονται και τόσο όσον αφορά την επικέντρωση για την αρχή της πρόνοιας και της πρόληψης και για τα αποτελέσματα και για τα θέματα μεθοδολογικά ε, εστιαζόμενοι σε αυτά και μια ολόκληρη σειρά θεμάτων που αφορούν την ε, ε, αναθεώρηση αυτού του πλαισίου. Σε σχέση με άλλα αποθέματα δεν υπήρχε χρόνος να καταδειχθεί ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι τα αποτελέσματα των μέτρων που αυτή τη στιγμή έχουν υιοθετηθεί για άλλα αποθέματα, όπως για παράδειγμα για τον Ξηφία ε, όσον αφορά και τον Ατλαντικό Βορρά και Νότο είναι από θέματα που έχουν ανακάμψει λόγω των μέτρων που υιοθετήθηκαν από την ΆΙΚΑΤ και βρίσκονται τώρα, θα έλεγε κανείς, ε, ε, σε καλύτερη κατάσταση από πλευράς υγείας αποθεμάτων. Καθώς επίσης και σε επίπεδα εκμετάλλευσης, λογικά επίπεδα θα έλεγα όπως επίσης και σε σχέση με το σπαθόψαρο ε, πρέπει να δούμε ότι σε σχέση με τις ε, ε, την κλίμακα στην οποία βρίσκεται είναι μεταξύ πράσινου και κίτρινου καθώς επίσης και τις επιπτώσεις των μέτρων διαχείρισης που είτε παρεμπόδισαν να επιδεινωθεί η κατάσταση αυτή, αυτών των αποθεμάτων και έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά είναι αποδεκτά επίπεδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση που δεν απάντησα σε αυτήν, αλλά νομίζω ότι κάλυψα τις παρεμβάσεις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ εσάς. Κύριε Ντάνερ, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Thank you, uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απλά σχετικά με τα θέματα που καλύφθηκαν. Πρώτα απ' όλα ως προς το προσφυγάκι. Δεν έδειξα όλα τα στοιχεία λόγω περιορισμού χρόνου. Η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι είχαμε μεγάλη αλία προσφυγακίου στην αρχή του 2001 στο 2002. Και πάλι η Ισλανδία, η Φερόες νήσι, η Νορβηγία και η Ρωσία αποφάσισαν ότι μπορούσαν ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς να αλλιεύουν. Δύο εκατομμύρια τόνων αυτού του είδους αλλιεύτηκαν μεταξύ 2003 και 2006, προτού τελικά επέλθει μια συμφωνία σχετικά με ε, την κατανομή των ελευμάτων. Το θέμα ήταν ότι άλλες ε, παράκτες χώρες πέραν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλίευαν ελεύθερα, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν όρια. Ενώ οι άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ότι ε, θα αλίευαν ανεξέλεγκτα. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Αλλά εκείνη την εποχή, ως εκπρόσωποι του κλάδου, νομίζαμε ότι δεν θα ξέφευγαν το πρόβλημα. Αυτό είναι. Ότι τελικά για την ανέθεση συμπεριφορά τους επιβραβεύθηκαν. Και πάλι εδώ το ίδιο βλέπουμε σε σχέση με το σκουμπρί. Διότι αν πάρετε το παράδειγμα που έχουμε στο προσφυγάκι, η Ισλανδία στο τέλος της δεκαετίας του 90 είχε το 2 ή 3% ε, ε, αλία στο προσφυγάκι. Τώρα έχει φτάσει στο 18-19%. Και το ίδιο συμβαίνει εδώ με το σκουμπρί. Γι' αυτό τονίζω συνέχεια αυτό το θέμα. Το τόνισα και στην παρουσίασή μου βεβαίως. Δεν κάλυψα όλες τις περιοχές. Δεν μίλησα για τα άλλα θέματα της οργάνωσης. Αλλά μας απασχολούν τα προβλήματα εκεί και κάτι πρέπει να γίνει. Και με τα χαράς διαπίστωσα ότι αρχίζει ο κόσμος να το βλέπει σοβαρά το θέμα και θα πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ, πρέπει να γίνει κάτι τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο. Γι' αυτό, ε, ακόμα και αν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αλίας έχουν περιορισμένο ρόλο, σίγουρα κάτι μπορούν να κάνουν. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουν ώστε κάτι να γίνει για να διατηρήσουμε την αηφορία ενός υγιούς αποθέματος. Και ε, ο ευρωπαϊκός στόλος και ο νευγικός στόλος εξαρτώνται από αυτό το είδος. Δεν πρέπει να αφήσουμε να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Έχουμε μια κακή εμπειρία με το προσφυγάκι, δεν πρέπει να επαναληφθεί. Ευχαριστώ πολύ για όσους έδειξαν αυτό το θέμα. Η κυρία Ζολή θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Ντόνα. Δεν... Ε, γνωρίζω τα θέματα, αλλά η δημοκρατική παράδοση της ε, Νορβηγίας και της Ισλανδίας ε, δεν θα το επέτρεπαν. Εκπλήσωμε που τα αλλιεύματα αυξήθηκαν τόσο πολύ. Και εσείς ξέρετε καλύτερα από εμά, αλλά ε, η μετανάστευση αυτού του είδους στο σκουμπρί άλλαξε. Το θέμα είναι πώς να χωρίσει κανείς τα αλλιεύματα, το αλλιεύμα. Υπάρχουν νέα δικαιώματα, διότι το σκουμπρί δεν πήγαινε εκεί. Μήπως αυτή είναι η εξήγηση ότι μετα... μετακινήθηκε το σκουμπρί προς αυτή την περιοχή. you, Ευχαριστώ. I'm glad you asked... Είμαι ευτυχής που θέσατε αυτό το ερώτημα, επειδή αυτό είναι πολύ εύστοχο ερώτημα. Δεν υπάρχει καμία, καμία δικαιολογία. Επειδή εφόσον επιδοκιμάζονται όσοι αλλιεύουν περισσότερο, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή μπορούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αλλιεύει 20 φορές παραπάνω από ό,τι έκανε. Διότι υπάρχει πάρα πολύ σκουμπρή στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι είδη τα οποία υπάρχουν και στα νορβηγικά ύδατα και στα ευρωπαϊκά ύδατα. Και ε, τα αποθέματα είναι απόλυτα υγιή. Υπάρχει σκουμπρί στην Ισλανδία και στις Φερόες νήσους, αλλά τα περισσότερα σκουμπριά βρίσκονται στα ευρωπαϊκά ύδατα. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν ότι εμείς θα αλλιεύουμε όσο μας αρέσει, επειδή τελικά θα υπάρξει υπεραλία. Πρέπει να υπάρχει τρόπος διαχείρισης των αλλιευμάτων. Υπάρχει ένα σύστημα, λοιπόν πρέπει να έχουν ευθύνη. Πρέπει να συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα προ τη διαχείριση των αποθεμάτων. Έχουν το δικαίωμα να λιεύουν ορισμένα, αλλά όχι τόσο πολύ. Από το 0 φτάσαν σε, σε 130.000 τόνους. Και στα πλαίσια της ΝΕΑΦ, εντάξει, αλλά όχι 130.000 τόνους, δεν το δέχομαι ε, σαν επιχείρημα. Επειδή το ψάρι βρίσκεται στα νερά σας, μπορείτε να ψαρεύετε όσο θέλετε τότε θα υπήρχε χάος σε κάθε αλληλευτική τακτική σε όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλω να σας πω ότι εγώ τα έχω δει και στην ΑΦΟ, ότι να υπάρχουν ε, συστάσεις, να υπάρχουν αποφάσεις για την Ισλανδία και τελικά να μην γίνεται αυτό που πρέπει, να κάνουν ό,τι θέλουν. Παρακαλώ κύριε Γκαράτ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις. Παρόλο που δεν απευθύνθηκε σε μένα η πρώτη της κυρίας Αντρές, με ρώτησε κατά πόσο ε, μπορούμε να προλάβουμε και να αποφύγουμε την παράνομη αλία του ερθρόπτερου τόνου. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει και μπορώ να σας εγγυθώ είναι ότι σε βαθμό που τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα φέτος και τον προηγούμενο, εφόσον έχουν εφαρμοστεί αυτά τα αυστηρά μέτρα, να ξέρετε ότι όποιοι πλειοκτήτες σκόπευαν να παραβούν τους κανονισμούς, η ζωή τους έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη τώρα. Και αυτό γιατί έγινε τεράστια προσπάθεια από όλες τις πλευρές. Και πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Και η ΚΑΤ το διαπιστώνει αυτό. Τώρα για την ερώτηση της κυρίας Λοβίν, κατά πόσο η ΚΑΤ θα έπρεπε να έχει περισσότερες δυνατότητες να επιβάλλει κυρώσεις. Ε, λοιπόν, λέω ότι ναι, θα έπρεπε και η ΚΑΤ και όλες οι περιφερειακές οργανώσεις, ώστε να αναγκάζουν τα κράτη-μέλη να τηρούν τους κανόνες. Όλοι οι φορείς, όλες οι πλευρές, όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν ε, στην αλληλευτική προσπάθεια. Τώρα, αν ε, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ένας νέος οργανισμός που να παίζει ρόλο συγκέντρωσης των περιφερειακών οργανώσεων αλίας και να τηρούν τους κανόνες και το δίκαιο της θάλασσας, κατά κάποιο τρόπο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια που έχουμε την αναθεώρηση της Συμφωνίας της Νέας Υόρκης, αυτό γίνεται από όλε τι πλευρέ Η κάθε περιφερειακή οργάνωση δηλαδή αναθεωρεί, βλέπει τι πρόοδου έχει πετύχει, βλέπει και τις αρνητικές πλευρές όπου υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια και ανάλογα προσαρμόζεται. Γίνεται λοιπόν αυτό. Γίνεται αυτή η αναθεώρηση. Και υπάρχει υποχρέωση αναθεώρησης των, του τρόπου λειτουργίας όλων των περιφερειακών οργανώσεων αλίας τώρα για ένα διεθνές ε, δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσας, μια τέτοια δυνατότητα είναι πάντα ανοιχτή. Τώρα πώς θα ολοκληρωθεί, αν γίνεται, αυτό είναι άλλη ιστορία. Τώρα για τις υπονάπτυξη χώρες, τις αναπτυσσόμενες, εμείς δεν είμαστε κατά βέβαια του να υπάρχουν τέτοιε δυνατότητες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρή κλίμακα σαλία που έχει άμεση σχέση με τα προϊόντα της χώρας και τη χώρα την ίδια. Το πρόβλημα είναι όταν οι αναπτυσσόμενες χώρες αυτό που θέλουν είναι να νοικιάζουν κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα αλίευσης από στόλους άλλων χωρών που τους έρχονται εκεί. Θα έπρεπε να υπάρχουν κανονικά ποσοστώσεις στις περιφερειακές οργανώσεις για να υπάρχει μια ισορροπία. Για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα αποθέματα. Τώρα ρωτήσατε κατά πόσο οι αλείς που παράνομα αλλιεύουν, αν μπορούν να συνεχίσουν να αλλιεύουν μέσα στις οργανώσεις περιφερειακής αλίας, ε, υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Αν τηρούνται έχει καλώς. Αν δεν τηρούνται πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Να τιμωρούνται γι' αυτό. Δυστυχώς, ε, μάλλον, ευτυχώς σε χώρες όπως είναι αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διαδικασίες που οδηγούν σε ποινές σε κυρώσεις. Αυτό που με ρωτάτε, εγώ θα σας το γύρναγα ως εξή. Αν πάει 30 χιλιόμετρα την ώρα παραπάνω πόσο πρέπει και η αστυνομία πιάσει το αυτοκίνητό σας, θα πάρετε βέβαια κάποια ποινή. Αν όμως είσαστε και μεθυσμένος, θα σας πάρει και το δίπλωμα, δεν θα ξαναοδηγήσετε ποτέ και θα καταλήξετε κατά πάσα πιθανότητα στη φυλακή. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αλία. Αν γίνει μια παράβαση, εντάξει, τρέχουσα ωραία, υπάρχουν κάποιες κυρώσεις. Αν ε, όμως γίνεται κάτι πολύ χοντρό, ε, δεν μπορεί κανείς να γενικεύσει δηλαδή και να σας δώσει μια γενικευμένη απάντηση. Ρωτήσατε ποια είναι η απόψή μου για τις σημαίες ευκαιρίες. Εγώ αντί να μιλήσω για σημαίες ευκαιρίες, θα μιλούσα για σημαίες που δεν τηρούν τους κανόνες. Γιατί η ιστορία των σημαίων ευκαιρίας είναι κάτι πολύ σχετικό. Ό,τι σημαία έχει ο καθένας είναι γιατί είναι μια καλή ευκαιρία για αυτόν. Οπότε άλλο αυτό και άλλο να έχει κανείς σημαία μιας χώρας η οποία επανειλημμένα παραβαίνει τους κανόνες και δεν δέχεται τους κανόνες ή τις αποφάσεις που έχουν ε, ληφθεί και τις διατάξεις που ισχύουν. Ορισμένοι εφοπλιστές ανά τον κόσμο αυτό κάνουν. Χρησιμοποιούν μια σημαία για να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχει μια διαφορά λοιπόν για μένα εδώ και σας τη λέω. Τώρα σε σχέση με την Greenpeace και με το αν υπήρξε παράνομη λίευση, από τη δικιά μας την πλευρά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γενικός γραμματέας της οργάνωσής μου, που είναι μία από τις οργανώσεις της Νομοσπονδίας. Δεν εκπροσωπώ όλες τις επιχειρήσεις, πάντως από τις πληροφορίες που έχω εγώ. Πρώτον, για το φυλάδιο της Greenpeace, που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες στην Κορούνια της Ισπανίας. Όπως συνήθως συμβαίνει, μπερδεύεται ε, ενημέρωση αντικειμενική, πραγματική και μη πραγματική. Κρίμα που ο κύριο Μουρών δεν είναι εδώ, γιατί εκείνο θα μπορούσε να σα παρουσιάσει καλύτερα τα θέματα. Πάντω, από τι πληροφορίε που έχω εγώ, αυτά τα οποία αναφέρονται δεν ισχύουν. Και μάλιστα είναι οι δικηγόροι τη οργάνωση που ασχολούνται να δούνε μήπω μπορούν να προσφύγουν κατά τη Greenpeace για αυτά που λέει στο φυλαδιό τη. Αυτό από μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά, φαντάζομαι ότι ξέρετε πω πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα ή την προπροηγούμενη, και μετά από τη δημοσίευση αυτού του φυλαδίου, μία ε, οργάνωση κατηγορήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με δικιά μας οργάνωση για παράβαση σε ύδατα κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρότειναν κυρώσεις 7,5 εκατομμύρια δολάρια για την παράβαση αυτή, για την παρανομία αυτή όπως ισχυρίζονται. Πρώτον ήταν μεγάλη έκπληξη για την επιχείρηση που δεν γνώριζε τα γεγονότα αυτά και δεύτερον τέθηκαν στη διάθεση των ΗΠΑ και της Ισπανίας που επίσης αναμειγνύεται στην υπόνοια παράβασης πήγανε στις Ηνωμένε Πολιτείε για να ενημερωθούν να ακούσουν τις εξηγήσει που είχαν να δώσουν οι Αμερικανοί και ενδεχομένως να αναλάβουν την ευθύνη εφόσον είχαν κάποια ευθύνη για την παράβαση του καπετάνιου του πλοίου, σύμφωνα με την κατηγορία. Η κατηγορία ήταν ότι πέταγαν πράγματα μέσα στα ύδατα των ΗΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλίευαν, σημαίνει ότι έριξαν στη θάλασσα ένα μηχάνημα, ένα εργαλείο αλίευσης, ώστε μια σημαδούρα ώστε σε 4, 5, 6 ώρες σιγά σιγά με τους μήνες παρασύρεται από τα νερά, μαζεύει, συγκεντρώνει μάλλον τον δόνο και αργότερα μπορεί να λιεύσει το πλοίο. Η επιχείρηση λοιπόν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευκρινιστεί η υπόθεση αυτή. Τέθηκε σε πειθαρχικό παράπτωμα ο καπετάνιος που είχε οδηγία να μην μπορεί να πετάξει αντικείμενα σε ύδατα για τα οποία δεν είχε άδεια και ανέλαβε την ευθύνη για το σφάλμα, για την αμέλεια αυτή του προσωπικού του, του πληρώματος. Από την αρχή όμως ξεκαθαρίστηκε ότι ούτε ένα τόνο δεν αλίευσαν. Σας είπα, πρόκειται για μία μέθοδο που μετά από μήνες μπορεί κανείς να αλλιεύσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Σύντομα θα μάθουμε οι συνομιλίες αυτές που θα έχουν καταλήξει. Σήμερα πάντως δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Όπως και να έχει το πράγμα όμως θέλω να σας πω ότι η επιχείρηση και το δημοσίευσε. Ανέλαβε την ευθύνη για το πλήρωμα και εξακολουθεί να επαναλαμβάνει την επιθυμία της να μπορεί να αλλιεύει όπου νόμιμα μπορεί να αλλιεύει. Ευχαριστούμε. Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, γι' αυτό θα ήθελα να κάνω ορισμένε παρατηρήσει και να σα δώσω ορισμένε ενδείξει σχετικά με το τι γίνεται τώρα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα που μα απασχολεί σήμερα. Δηλαδή, η μεταρρύθμιση τη εξωτερική διάσταση τη κοινή ελευθερική πολιτική. Καταρχήν, νομίζω ότι μιλήσαμε για τον ερυθρό τόνο, όπω εξηγείται συνήθως όταν μιλάμε για τα θέματα των οργανώσεων και ορθά ο ερυθρός τόνος αποτελεί πολύ μικρό ποσοστό των ε, ειδών που αλλιεύονται από τις οργανώσεις. Νομίζω ότι αυτό το είδος ήταν προβληματικό. Και επέστησε την προσοχή του κοινού και των πολιτικών και τώρα, αν θέλετε, είναι το, ε, δέντρο που κρύβει ε, το δάσος το θέμα είναι πολύ ευρύτερο και δεν περιορίζεται εκεί. Υπάρχουν και άλλα είδη, όχι μόνο ο ερυθρό των Διότι δεν είναι μόνο η ΚΑΤ η οποία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο ε, στη διαχείριση ε, αυτών των ειδών. Δεύτερη προκαταρκή παρατήρηση. Μιλήσαμε για τη Συμφωνία της Νέας Υόρκης που έγινε πράγματι εκείνη η οποία το 1995 ανέθεσε ε, μεγάλη σημασία ε, στι περιφερειακέ οργανώσει. Ε, και κατόπιν ορισμένε οργανώσει δημιουργήθηκαν. Και επίση αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα, διότι πολλέ οργανώσει Αλίας είναι νέε, είναι νέε οργανώσει μικρή ηλικία. Συνεπώς μπορούν να κάνουν πολύ πρόοδο ακόμα και γι' αυτό α του δώσουμε χρόνο, ώστε να μπορέσουν να διαδραματίσουν πλήρως το ρόλο τους και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω, έχει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω της παρουσίας του στόλου της σε όλο τον κόσμο, λόγω των επενδύσεων, λόγω της παρουσίας της στις οργανώσεις αυτές και λόγω του μεγάλου ρόλου της ε, αγοράς μας στην εισαγωγή αληφτικών ειδών και ω προ τον διεθνή ρόλο που θέλουμε εμεί να διαδραματίσουμε για την προστασία τη βιοπικιλότητα. Όταν μιλάμε για τι οργανώσει, δεν μιλάμε για τη γραμματεία που διαχειρίζεται τα πράγματα, αλλά οι αποφάσει λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σημαντικό παράγον σε πολλέ οργανώσει και πιστεύω έχει ιδιαίτερη ευθύνη για να βελτιώσει την επίδοση αυτών των οργανώσεων. Τώρα, θα ήθελα να σας διαβιβάσω ορισμένε σκέψεις σχετικά με την αναμόρφωση αυτών των οργανώσεων, των προεδριακών οργανώσεων. Και νομίζω ότι ε, ε, συμφωνούμε με τα σχόλια, πρώτα απ' όλα, το θέμα της επιστημονικής άποψης. Και το θέμα της ποιότητας αυτών των επιστημών απόψεων είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να υπάρχει καλή διαχείριση αυτών των οργανώσεων. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να είναι ποιοτικέ εργασίες που γίνονται, το οποίο σημαίνει επενδύσεις επενδύσεις, ανθρώπινους πόρους, σε χρήματα, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να συμβάλλει ε, στις επιστημονικές εργασίες που γίνονται και κατόπιν οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται να είναι σύμφωνες με τις επιστημονικές απόψεις. Πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζει μία από τις βασικές αρχές της κοινής ελευθερικής πολιτικής. Δεύτερο στοιχείο είναι το θέμα να γίνονται σεβαστές υποχρεώσεις, compliance στα αγγλικά. Πολλές από αυτές τις οργανώσεις έκαναν αμαρτίες, υπό την έννοια ότι η, η, η, η υλοποίηση των μέτρων δεν ήταν ικανοποιητική. Γι' αυτό σε πολλές από αυτές ε, τις οργανώσεις και η ΚΑΤ προσπάθησε, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε άρδιν τον τρόπο με τον οποίο τηρούνται οι υποχρεώσεις. Πώς ε, γίνεται η επιτήρηση, πώς συζητούνται, πώς γίνεται διόρθωση των μέτρων και αν παραστεί ανάγκη και αν υπάρχει άλλος τρόπος να προβλεφθεί επιβολή κυρώσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για να μπορέσουμε να καταλήξουμε εκεί φυσικά πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα ελέγχου πρόκειται για, τον, για την ευθύνη ε, της χώρας που έχει τη σημαία ή την, το λιμάνι ή και το θέμα της χώρας που είναι υπεύθυνη για την αγορά αυτό έγινε για να αντιμετωπιστεί η υπεραλία. Γι' αυτό παροτρύνονται μεγάλε αλληλευτικέ χώρε να υιοθετήσουν αντίστοιχε νομοθεσίε και μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ε, την παράνομη αλία. Τώρα, ω προ το θέμα τη στήριξη των υποχρεώσεων, αυτό το θέμα είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι ουσιαστικό. Διότι είναι περιττό να υιοθετούμε μέτρα εάν κατόπιν δεν εφαρμόζονται. Κατόπιν έχουμε το θέμα της διαχείρισης της ε, ε ικανότητας ε, του στόλου υπάρχει σε ορισμένε περιπτώσει υπερβολική ε, χρήση του στόλου και να φόκειται στι αναπτυσσόμενε χώρε όπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει προσπάθεια. Αλλά δεν πρέπει αυτή η προσπάθεια να είναι περιττή. Διότι τι να κάνουμε ε, ε, το, το στόλο, να τον περιορίζουμε, αν άλλοι τον αυξάνουν το στόλο του. Είναι πολύ ευαίσθητο. Το θέμα είναι μπορούμε να περιορίζουμε το στόλο μα ώστε να μην είναι υπερβολικό και κατόπιν οι θεμητέ προσδοκίε των αναπτυσσομένων χωρών ώστε να συμμετέχουν περισσότερο στην αλία ή τουλάχιστον στα ποιο που απορρέουν από αυτή την αλία. Τώρα έρχομαι στην τέταρτη παρατηρήσή μου. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών. Αλληλευτική πολιτική, αλλά και εμπορική πολιτική, συνοχή με την περιβαλλοντική πολιτική και συνοχή με την αναπτυξιακή πολιτική. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής Αλλίας και Ανάπτυξης. Το θέμα αυτής της συνοχής μεταξύ Αλλίας και Ανάπτυξης είναι κεντρικό σε πολλέ από αυτέ τι οργανώσεις, οι περισσότερε συμμετέχουσες χώρες είναι αναπτυσσόμενε. Η πρώτη πρόκληση είναι ακριβώ πώ θα συμμετέχουν πραγματικά στι εργασίε αυτών των επιτροπών. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση τακτικά χρηματοδοτεί τη συμμετοχή αυτών των χωρών και των επιστημόνων του στι εργασίε αυτών των οργανώσεων. Αυτό το θέμα είναι πολύ απλό, αλλά είναι πολύ σημαντικό, ώστε να μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν στι εξελίξει. Τέλο, ε, το θέμα τη τεχνική βοήθεια, και τη ενίσχυση των ικανοτήτων του πώς μπορεί να ενισχυθεί η ικανότητά τους να ελέγχουν την αλία ή και να αναλαμβάνουν επιστημονικέ έρευνε προτού να είναι ικανέ αυτέ οι χώρε να διαχειρίζονται το στόλο του, το στόλο των τρίτων χωρών που αλλιεύουν στα νερά του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που καλύπτεται κυρίω μέσω των ε, συμπράξεων αλεία που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο στοιχείο. Το θέμα ε, του μεριδίου τους ε, σε αυτό το γλυκό που θα λέγαμε. Δηλαδή, τι μερίδα θα πάρουν ε, αυτές οι χώρες. Για ιστορικούς λόγους, το μερίδιό τους περιορίζεται. Δηλαδή, οι χώρες τους, όπως οι εταίρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Αλλά με την βάση των ετών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να τους δώσει χώρο, ώστε ε, αυτές οι, χώρες, να μπορέσουν να συμμετέχουν περισσότερο στην Αλία. Μιλούσαμε για την ΙΚΑΤ. Πέρσι στην ΙΚΑΤ ακριβώ τα μέτρα ε, για τον ξηφία του Νοτιού Ατλαντικού αναθεωρήθηκαν και δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει το δικό τη το μερίδιο, την ποσόστοσή τη δηλαδή, και να αφήσει μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτέ τι χώρε. Εκεί λοιπόν κάνουμε προσπάθειε κοστίζει για τον ευρωπαϊκό στόλο, κοστίζει για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αλλά ανταποκρίνεται στην ιδέα που έχουμε για την αναπτυξιακή μα πολιτική. Τέλος, ε, τελευταία παρατήρηση, όπω σα έλεγα, το θέμα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο στόλο, αλλά γενικότερα περιορίζεται στο θέμα των ωφελών. Δηλαδή, ότι μπορούμε να ωφεληθούμε από τον περιορισμό ε, ε, του, του στόλου, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις ε, να υπάρχουν μεταπητικές βιομηχανίες, ε, κονσερβοποιίες. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα περιλάβουμε στην πολιτική αλίας και στην πολιτική ανάπτυξη, ώστε να έχουμε μια συνεκτική πολιτική που θα εξασφαλίζει τη ισορροπία μεταξύ των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και το όραμά μας, το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτός ο θεματολογικός γύρος, ε, αυτή η κατηγορία. Φτάσαμε 4,5. πρέπει να δούμε τις διμερείς συμφωνίες ε, αλληλείας. Ε. σε σχέση με τις χώρες του Νότου. Είναι μια πολιτική πρωτοβουλία με την πολιτική ανάπτυξη η κυρία Ζολή είναι παρούσα και της Επιτροπής Αλίας. Το ίμιση των που έχουν προσκληθεί είναι από την Επιτροπή Ανάπτυξης, το άλλο ίμιση από την Επιτροπή Αλληλείας. Θα παρέμβουν και ευρωβουλευτές της Επιτροπής Αλληλείας και της Επιτροπής Ανάπτυξης και η κυρία Ζολή θα δίνει τον λόγο στην, στα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, εγώ στα μέλη της Επιτροπής Αλίας και έτσι θα εναλλασσόμαστε τα μέλη των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών ώστε να διασφαλίσουμε ότι και οι δύο επιτροπέ και τα, οι μέλη αμφωτέρων των επιτροπών θα μπορέσουν να παρέμβουν και την κυρία Μιλάτ που μας ε, καλωσορίζει, καλωσορίζω που μας συνοδεύει στις εργασίες μας, ε, καλωσορίζω και από πλευράς της Επιτροπής ε, θα υπάρξει ενημέρωση για τις προόδους που έχουν σημειωθεί σε αυτό το επίπεδο. Καλωσορίζω την κυρία Ζολή και δίνω τον λόγο για να πέντε λεπτά, ώστε στη συνέχεια να επικεντρωθούμε στη συζήτηση έχετε τον λόγο για να μπορέσετε να παρέμβετε ενώπιον των μελών της Επιτροπής Αλίας και Ανάπτυξη, Ανάπτυξης και Αλίας καλύτερα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ευτυχής που γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ, επειδή η Επιτροπή Ανάπτυξης παρέχει συμβουλές, απόψεις για τις αλληλευτικές συμφωνίες και μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι τις ονομάζουμε συμπράξεις και έχουν ένα αναπτυξιακό σκέλος. Δεν βλέπω ότι μέσω αυτών των συμφωνιών πραγματοποιούμε αναπτυξιακό έργο. Είδαμε σήμερα τη Συμφωνία Αλία Σολομού και αυτό και αυτή είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου. Τους δίνουμε δηλαδή 65 δολάρια τον τόνο. to Το είναι σωστό, είναι δίκαιο. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Και από ε, στο ε, δεδομένο ότι το άρθρο 208 της Συνδίκη Λισαβόνα λέει ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ όλων των εξωτερικών πολιτικών τη Ένωσης, πιστεύουμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης ότι οι αλληλευτικές συμφωνίες ίσως δεν θα πρέπει να συνδέονται με την ανάπτυξη και ότι αφενός θα έχουμε την ανάπτυξη και αφετέρου θα έχουμε τις ε, πραγματικά εμπορικές αλληλευτικές συμφωνίες. Επίσης, έχω και άλλη μια παρατήρηση. Στην προετοιμασία αυτής της κοινή συνάντησης, η αρχική ιδέα να υπάρχει εμπειρογνώμονας από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, αυτό το είπε ένας σύμβουλος που έκανε την ανεξάρτητη αξιολόγηση ε, των συμπράξεων αλίας για την Επιτροπή. Στις αρχές Μαΐου συμφωνήσαμε να παραβρεθούμε υπό την περιπτώση ότι θα συμφωνήσει και η Επιτροπή. Αυτό ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Συνεπώς, ε, θα μπορούσε και η εμπιστευτικότητα να τηρηθεί. Κατόπιν ζητήσαμε στην επιστροπή, η οποία δίστασε επί τρει εβδομάδε, προτού μα πει ότι δεν θα ήταν ευστοχό για το Συμβούλο να είναι παρόν. Η Επιτροπή είπε ότι ήθελε μόνη να παρουσιάσει το θέμα, το οποίο όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κατόπιν εξεπλάγημεν όταν ε, πριν από μια εβδομάδα μας είπε ο Σύμβουλος ότι άλλαξε γνώμη ε, και θα ήθελε να συμμετάσχει. Ενώ εκτιμούμε την ξαφνική αλλαγή από πλευράς Επιτροπής, ε, ήταν πολύ αργά. Εν τω είχαμε ε, καλέσει κάποιο Νορβηγό ε, εμπειρογνώμονα της Αλίας. Η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, θα καλέσει έναν ειδικό για την ανάπτυξη να πει τη γνώμη του. Εν τω μεταξύ, θα θέλαμε να μας πει η Επιτροπή κατά πόσο η Γενική Αξιολόγηση της Συμφωνίας θεωρείται ότι ανήκει στο δημόσιο χώρο. Well, we have been sent the general evaluation of σε Σεστάλη η γενική αξιολόγηση τη αλληλευτική σύμπραξη που διεξήγαγε ο Σύμβουλος και ειλικρινά δεν βλέπω γιατί ανησυχούσε η Επιτροπή. Δεν υπήρχε τίποτα το αμφιλεγόμενο ή το ε, δύσκολο. Ε, τα πορίσματα είναι τα εξή. Οι πληρωμέ για αυτέ τι συμφωνίες είναι 18% του συνολικού προπολογισμού αλίας και προβλέπουν πρόσβαση για πάνω από 300 ε, πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τα δύο τρίτα από την Ισπανία. Δηλαδή 14% ε, του συνολικού ευρωπαϊκού στόλου. Οι, τα ε, αντιστοιχούν σε 400.000 τόνους ετησίως, 8% της συνολικής ευρωπαϊκής αλίας. Αλλά το 3% μόνο της συνολικής κατανάλωσης. Επίσης, ορισμένα από αυτά στάλησαν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα δύο τρίτα κατανεμήθηκαν στις τρίτες χώρες με τις οποίες είχαμε συμφωνία. Ορισμένες συμφωνίες δημιουργούν 1.700 εργασίες, κυρίως για την Ισπανία και τη Γαλλία και 4.300 εργασίες για τρίτες χώρες. Όσον αφορά τις πληρωμές στις τρίτες χώρες, οι κοινοτικές πληρωμές είναι γενναιόδορες σε σχέση με ε, τα αλλιεύματα. Η αξιολόγηση περιορίζεται σε στατιστικά στοιχεία. Λιγότερο λέγονται για τη συνεισφορά των συμπράξεων στην αηφόρο ανάπτυξη του αληφτικού κλάδου ή στη βελτίωση της διακυβέρνησης στις χώρες εταίρους. Ε, ωστόσο έγιναν λίγες παρατηρήσεις. Η καταπολέμηση ε, ορισμένων αλλιευμάτων όπως ε, για τη Βόρεια και Δυτική Αφρική και ορισμένες πλευρές του Δικού Κενού, κατά τα λοιπά, ε, αυτά τα λιεύματα είναι περιορισμένα για την παράνομη αλία του γιογιό, με το γιογιό. Επίσης, ε, αυτή η αλία αφορά ορισμένους, ορισμένες ζώνες. Όσον αφορά τις επιστημονικές έρευνες, δεν είναι επαρκής οι κανόνες βελτιώνονται στις τρίτες χώρες, κυρίως εκείνε οι οποίες έχουν οικονομικές συμφωνίες. Ε, οι χώρες που δεν έχουν αρκετέ συμφωνίε ε, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσει εξαγωγών τη ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά ε, τις μεταρρυθμίσει, η αξιολόγηση υπογραμμίζεται εξή. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει διαχωρισμό μεταξύ του των αλληλευμάτων ε, αυτών των χωρών και των τρίτων χωρών και η, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διαπραγματευτεί με τρίτη χώρα, θεσπίζοντας ελάχιστες συνθήκες ε, για ε, τη λειτουργία των αλληλευτικών πλοίων. Η υποστήριξη της ανάπτυξης διαχωρίζεται από την πρόσβαση στην αλληλεία και βασίζεται στον προσδιορισμό των αναγκών της ανάπτυξης των τρίτων χωρών με την επιλογή να παρασχεθεί βαθμιαία υποστήριξη ανάλογα με την πρόοδο που επιτελείται. Ε, επίσης, περιφερειακές λύσεις με την υποστήριξη των περιφερειακών αρμοδίων οργανώσεων για την αντιμετώπιση των κοινών ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι παράκτιες χώρες που βρίσκονται στην περιοχή η Επιτροπή Ανάπτυξης ενδιαφέρεται και για αυτές τις δύο προσεγγίσεις και μάλιστα καλέσαμε έναν εμπειρογνώμονα από τον Οργανισμό Αλίας του Ειρηνικού να μας εξηγήσει την περιφερειακή τους προσέγγιση στις συμφωνίες για τον τόνο, αλλά βρίσκονται όλοι στην Αυστραλία αυτή την εβδομάδα σε μια διεθνή συνάντηση για τον τόνο και δεν μπορούν να παραβρεθούν. Η Επιτροπή Ανάπτυξη ε, προτίθεται να τους καλέσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Είμαι πολύ ευτυχής που θα δώσω τώρα το λόγο σε έναν παλιό συνάδελφο. First uh, okay, so, well, that, this was my introductory... Ήταν, ε, αυτές ήταν οι εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Θα δώσω το λόγο σε εσάς τώρα. Ναι, θέλω κι εγώ να πω ότι δεν θέλουμε πολεμική εδώ, αλλά αυτές οι ελευτικές συμφωνίες ακούμε ότι δεν ε, παίζουν το ρόλο τους στον αναπτυξιακό. Ναι, αλλά ποια είναι η γραμμή στον προπολογισμό που έχουμε για όλες τις ελευτικές συμφωνίες, 160 εκατομμύρια ευρώ. Με τα χρήματα αυτά γίνονται πάρα πολλά για την ανάπτυξη ναι. στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και φυσικά και θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα αυτά, είναι ψίχουλα. Δεν είναι δυνατόν να βάλουμε και την ανάπτυξη με τα χρήματα αυτά. Έτσι κι είναι δύσκολο. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στους δύο προσκεκλημένους της Επιτροπής Αλίας και μετά η κυρία Ζολή θα δώσει το λόγο στους άλλους δύο προσκεκλημένους, προσκεκλημένους της Επιτροπής Ανάπτυξης. Για 10 λεπτά λοιπόν, καταρχήν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μουριέλ, που είναι ο πρόεδρος της Αναμάρ, που είναι η Ισπανική Ένωση των ε, Σκαφών, των Αλληλευτικών για τα Οστρακόδερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο Επιτροπή Ελίας όσο και Επιτροπή Ανάπτυξης, για να συμμετάσχω σε αυτήν τη δημόσια κρέωση για την εξωτερική διάσταση της μεταρρύθμισης της κοινή ελευτικής πολιτικής και ιδιαίτερα όσον αφορά τις συμφωνίες σύνδεσης με τις χώρες του Νότου. Η παρέμβασή μου έχει σαν στόχο να εξηγήσω στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πόσο μεγάλη σημασία έχει το κοινοτικό στόλο και για την αλίευση βεθοπελαγικών ειδών η συνέχιση των συμφωνιών αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Το ότι έχετε 10 λεπτά, λέει η Πρόεδρο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάτε ακόμα πιο γρήγορα, γιατί πρέπει και να σα μεταφράσουν οι διερμηνεί. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο μιλητή. Είμαι πλειοκτήτη, εφοπλιστή και έχω μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, συγκεκριμένα η μητέρα μου, τα τρία μου και εγώ. Έχουμε λοιπόν μηχανότρατε, ε, ψυγεία, τέσσερις ισπανικής ε, σημαία και πέντε από τη Σενεγάλη και αλλιεύουμε στην Μαυριτανία και στην Γινέα Μπισάου, οστρακόδερα και κεφαλόποδα. Είμαστε μια οργάνωση από το 1977. Έχουμε την έδρα μας στην Ουέλβα και η δραστηριότητά μας είναι πολύ σημαντική για την ε, περιοχή. Η Αναμάρα συμμετέχει στην ε, Ισπανική Νομοσπονδία Ελίας με στόλους για βυθοπελαγικά είδη, κεφαλόποδα, μερλούκιο έχουμε παραγαδιάρικα στην οργάνωσή μας. Εδώ θα αναφερθώ λίγο στην πράσινη βίβλο που έλεγε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την συνοχή όλων των στοιχείων της κοινή αλληλευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδιαίτερα σημασία έχει η αναπτυξιακή πολιτική και το περιβάλλον. Εδώ θα προσθέσω και έρευνα και υγεία. Γιατί είναι και αυτά πτυχές πολύ σημαντικές, όπως και το εμπόριο, πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη. Είμαι, όπως σας είπα, εφοπλιστής και έτσι έχω μπορέσει να δω από πρώτο χέρι τι έγινε με την εξαφάνιση παραδοσιακών συμφωνιών, όπως για παράδειγμα με την Αγκόλα, τη Σενεγάλη, τη Μοζαμβίκη, όπως επίσης και τι έγινε όταν εξαφανίστηκε το ειδικό μας καθεστώς στις συμφωνίες με το Μαρόκο, την Καμπόν ή την ε, Ακτή Χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Έτσι λοιπόν ο στόλος της οργάνωσής μας, της Άννα από 200 σκάφη που είχαμε με ισπανική σημαία το 80-90, φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, μόνο με 48. Ο κοινοτικό στόλος αλείβει κυρίως στην Μαυριτανία και την Κινέα Μπισάο βάσει συμφωνιών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες αυτές. Επίσης, ελεύουμε και στην Αγγόλα και στο Κονγκό με ειδικέ προσωρινές συμφωνίες. Παρά τις επικρίσεις που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια, ε, δυστυχώς έχουμε δει ότι έχει αφήσει τεράστιο κενό πίσω του ο αλλιευτικός ε, κοινοτικός ε, στόλος σε ύδατα τρίτων χωρών, που καλύφθηκε όμως από σκάφη τρίτων χωρών, αναδιόμενων αλλιευτικών δυνάμεων που δεν τηρούν τους κανόνες, ούτε υγιεινείς, ούτε εργασιακούς κανόνες, ούτε για το περιβάλλον και τι έχει συμβεί με τους πόρους τους αλλιευτικούς στις περιοχές αυτές. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ για να σας κάνω να καταλάβετε ότι παρόλο που οι συμφωνίες αυτές καθ' άλλο τέλειε είναι και θα έπρεπε πολλά σημεία να αλλάξουν, παρόλα αυτά το ωφέλη για τις δύο πλευρές που υπογράφουν τέτοιες συμφωνίες είναι πολύ μεγάλα. Έτσι λοιπόν εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2004 όπου σαφώς αναφέρεται η βούληση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν με τις αλληλευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, κάτι το οποίο να αποτελεί στοιχείο κλειδί τη όποια κοινή ελευθερικής πολιτικής. Πράγματι, οι Ελευτικέ συμφωνίες αποτελούν ένα πολύ ε, σημαντικό νομοθετικό μέσο που έχει στη διάθεσή του ο κοινοτικό ελευθερικός στόλο για να μπορεί να λιεύει σε ύδατα τρίτων χωρών με ωφέλη, όχι μόνο οικονομικά, και μάλιστα ωφέλη και για τις δύο πλευρές και η Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να λιεύει εκεί, αλλά και ωφέλη για τις ε, χώρες ε, ε, στον οποίο τα ύδατα αλλιεύουμε. Οι χώρες αυτές λοιπόν έχουν κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρόνως αυξάνονται οι θέσεις απασχόλησης εκεί, η εμπορία, ασχολούνται με την μεταποίηση, με την επισκευή σκαφών επίσης, έχουν ωφέλη από τις λιμανικές δραστηριότητες ε, και όλες οι δραστηριότητες στα λιμάνια υποφελούνται, τα τελωνία, μετανάστευση κλπ. Θέσεις απασχόλησης, πολύ σημαντικό. Και καταπολέμηση τις παράνομες αλλιές επίσης. Όσον αφορά τώρα τις συμφωνίες στα πλαίσια ε, αυτά, ιδιαίτερα για τη Μαυριτανία, την Κινέα Βυσάου και το Μαρόκο, πρέπει να σας πω ότι λήγουν οι σχετικές συμφωνίες. Εκείνη με το Μαρόκο το Φεβρουάριο του 2011, με την Γινέα Μπισάου τον Ιούνιο του 2011 και με τη Μαυριτανία τον Ιούλιο του 2012. Αυτές οι τρεις χώρες μάλιστα, πέρα από το ότι έχουν ωφέλη, όπως αυτά που σας ανέφερα πριν, έχουν και οικονομικά ανταλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο βοηθάει πολύ τους εθνικούς τους προπολογισμού. Όπως έλεγε πριν και η πρόεδρος της Επιτροπής, η οικονομική ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των συμφωνιών αυτών έχει μειωθεί από 250 εκατομμύρια σε 160 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια. Έλεγα στην αρχή ότι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι κάποιες πτυχές των αλληλευτικών αυτών συμφωνιών πρέπει να βελτιωθούν και γι' αυτό πρέπει από κοινού σε στενή συνεργασία με τις εθνικές ε, κυβερνήσεις και τις κοινοτικές αρχές να συνεργαστούμε. Όπως επίσης και με την επιστημονική κοινότητα και τους αλείς. Έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερα, καλύτερες προδιαγραφές για τις επόμενες συμφωνίες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Μαρόκο μπορούν να βελτιωθούν οι λευτικές συμφωνίες, ώστε ο αλλιευτικός στόλος από την Ανταλουσία να μπορεί ελεύθερα να λιεύει στην περιοχή εκεί με συνεργασία με τις αρχές του Μαρόκο. Χρειάζεται ανανέωση της συμφωνίας με το Μαρόκο με βελτιώσεις. Στην περίπτωση τώρα με την Μαυριτανία και την Γινέα Πισάου, όπου χρησιμοποιούνται πλήρως οι διατάξεις των αλληλευτικών συμφωνιών, και εδώ μπορούμε να βελτιώσουμε τις συμφωνίες αυτές. Είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε το ίδιο επίπεδο ελέγχου για του τόλου που αλλιεύουν σε ύδατα χωρών. Επίση, για το πρωτόκολλο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για μα αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε να θεσπιστούν οι αναγκαίοι μηχανισμοί για να διασφαλίσουμε ότι ένα μέρο του αντισταθμίσματος οικονομικού που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει για τη συνεργασία και ανάπτυξη. Το μικρόφωνο του ομιλητή είχε βλάβει και να βοηθήσει για την αηφορία στην αλληλεία και για να βελτιωθεί η προσπάθεια σε σχέση με τις χώρες αυτές. Σε σχέση με το αντιστάθμισμα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ποιο θα πρέπει να είναι το αντιστάθμισμα που θα οδηγεί στη, οδηγείται στην ε, συνεργασία και την ανάπτυξη της χώρας και ποιο θα είναι το αντιστάθμισμα το οποίο θα αφορά τους πόρους. Θεωρούμε ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη που προβλέπεται από τη Συμφωνία πρέπει να ε, χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Και αντίστοιχα θεωρούμε ότι οι εφοπλιστές ε, θα έπρεπε να επομίζονται μόνο την αντιστάθμιση της αξίας στην πρόσβαση των αλλιευμάτων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη όμως το υψηλό κόστος που πρέπει να επομίζονται οι εφοπλιστές για να ασκούν αλλιευτικές δραστηριότητες σε τρίτες χώρες, μακριά από την έδρα τους, με το κόστος της περατζάδας, της διαδρομής αυτής και όλα τα σύναφη για να καθορίσουμε τη συνεισφορά των εφοπλιστών είναι αναγκαίο να καθορίσουμε την δίκαια τιμή για την πρόσβαση στους αλλιευτικούς πόρους στα ύδατα των τρίτων χωρών. Αυτό το κριτήριο όσον αφορά την κατανομή των αντισταθμιστικών αυτών ωφελών θα πρέπει σε όλες τις συμφωνίες ε, να είναι ίσο και δίκαια, μερές και δίκαιο. Από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφέρουμε ότι σε σχέση με τις συμφωνίες ε, που αφορούν ε, τις ε, ιδιαιτερότητες τρίτων χωρών, αν και κάποιες στιγμές ε, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα για τις αλλιευτικές εταιρείες που ασκούν εκεί δραστηριότητες, για παράδειγμα σε σχέση με την κατάσταση λόγω απαγορευμένων δραστηριοτήτων σε κάποιες ζώνες είναι το μόνο νομικό ε, μέσο το οποίο έχουν ε, οι κοινοτικά εμπλεκόμενοι για να μπορέσουν να προασπίσουν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους ε, μέσα σε ένα συναφές πλαίσιο. Γι' αυτό πρέπει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα ώστε να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια που να στοχεύει στο να διασφαλίζει τη σωστή υλοποίηση των όσων θεσπίζονται στα πρωτόκολλα. Έτσι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος της Μικτής Επιτροπής, Μικτής Επιτροπής ως ε, φόρουμ που θα δίνει συνέχεια στην εφαρμογή των συμφωνιών, όπου ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, εμπλεκομένων μερών, θα δίνει τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να πρικοδοτηθεί η Γενική Διεύθυνση όσον αφορά την, ε, την Επιτροπή για την Αλληλεία να έχει το μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό και το μεγαλύτερο ε, υλικό δυναμικό για να μπορέσει να προωθήσει αυτούς τους στόχους βασιζόμενοι στον αλληλευτικό τομέα και τα, την πείρα που έχει καθώς επίσης και την βοήθεια την επιστημονική ώστε να μπορούν να διασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ της αηφορίας, της οικονομικής ε, αλλιευτικής δράσης και των, της διατήρησης και διασφάλισης των αλλιευμάτων. Εν τέλει θα ήθελα να αναφερθώ ε, ξεχωριστά στην ρήτρα ε, αποκλειστικότητας και στην ανάγκη να εμπλέκεται και να είναι κατανοητό αυτό σε σχέση με τον αλληλευτικό τομέα. Θεωρούμε ότι αυτή η ρήτρα υπό συγκεκριμένε προϋποθέσεις μπορεί να είναι δικαιολογημένη όπου δεν είναι σε σωστή κατάσταση τα αλλιεύματα μιας χώρας. Όμως πρέπει να υπάρχει και κοινή λογική όταν έρχεται η στιγμή να εφαρμοστεί σε διαφορετικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό ολοκληρώνοντα να τονίσουμε ότι ο στόχος, οι στόλοι που αλλιεύουν μέσω των ε, ε, μεικτών συμφωνιών, κεφαλόποδα για παράδειγμα, θα πρέπει να έχουν την έγκριση της συμφωνίας αυτής όπως και με τη Μαυριτανία και την Γινέα Μπισάου. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για τον κοινοτικό στόλο η υπογραφή των συμφωνιών με την Σενεγάλη με αντίστοιχα σκάφη που θα, 30 ε, που θα δραστηριοποιούνται εκεί ή με την Αγγόλα για τη δραστηριοποίηση 70 σκαφών. Και πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνοντα να καταβάλει την μέγιστη προσπάθεια για να μπορέσει αυτή η δραστηριότητα να διασφαλιστεί. Από την άλλη πλευρά όλοι δείχνουν και θέλουμε να πούμε ότι είμαστε απόλυτα πρόθυμοι να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στην αναζήτηση των ε, αναγκαίων και σωστών μέσων για να διασφαλιστεί η πολιτική αυτή αυτή για την αλία και να βελτιωθεί η απόδοσή της. Κύριε Προβουλευτέ, δεν θα πρέπει να επιτραπεί να χαθεί μια τέτοια θεμελιώδης δραστηριότητα κοινωνικά, οικονομικά ε, από πλευρά ζωνών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό την αλία όπως στη Γαλλικία, στα Κανάρια νησιά ή στην Ανδαλουσία ή και σε άλλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που μεγάλες θυσίε συνεπαγόταν η πολιτική αυτή και πολλές οικογένειες εξαρτώνται από αυτή τη δραστηριότητα ώστε να μπορέσουν να διασφαλίσουν τη διαβίωσή τους. Μπορείτε να, δείτε, να πάρετε και ένα αντίτυπο στα αγγλικά και στα ισπανικά του λόγου μου πίσω εκεί στο βάθος στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος και η κυρία Μπερτής Κορές που είναι η συντονίστρια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 Θα δώσω τώρα στο, το λόγο στον κύριο Αχμέτ ε, Σερίφ, που είναι πρόεδρος της ΠΕΣΚΟΠΣ από τον Νουακτσότ της Μαυριτανίας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση αυτή για την πράσινη βίβλο αποτελεί ένα παράδειγμα χρηστής διακυβέρνησης Βούληση για διαφάνεια από όλε τι πλευρέ. Η διαβούλευση με όλες τις πλευρές είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα καταλήξουμε σε καλά μέτρα, τα οποία να τεθούν και σε εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, παρά τη τεράστια πρόκληση που αποτελούν τα πέντε διαρθρωτικά προβλήματα της κοινή ελευτικής πολιτικής, παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξο όσον αφορά την διαδικασία αυτή, η οποία θα έπρεπε να μας επιτρέψει να καταλήξουμε στη, στο όραμα για την Ευρωπαϊκή Αλία του 2020. Εξάλλου είναι ένα όραμα που έχουν και οι αλίες της Δυτικής Αφρικής. Οι προκλήσεις μάλιστα στη δικιά μας την πλευρά είναι πολύ μεγαλύτερες. Και γι' αυτό και χρειαζόμαστε βοήθεια από τις πλούσιες χώρες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα. Οι συμφωνίες αλληλευτικής σύμπραξης είναι συμφωνίες από τις οποίες δεν επωφελείται μόνο η Δυτική Αφρική. Παράδειγμα, ναι, έχουμε τα περισσότερα ευρωπαϊκά ε, σκάφη και τα τελευταία χρόνια υιοθετήσαμε πολλές τομιακές πολιτικές όσον αφορά την αηφόρο εκμετάλλευση των πόρων με ωφέλη για την εθνική οικονομία. Όμως, η πίεση που είχαμε τελευταία για περισσότερα έσοδα οδήγησε σε μασική πώληση αδειών αλληλευτικών σε ξένους στόλους με αποτέλεσμα να ε, έχουμε μεγαλύτερη μείωση των ε, αποθεμάτων, κάτι το οποίο έχουν υπογραμμίσει ομάδες εργασίας και της ΚΟΠΑΣΕ και ομάδες εργασίας επιστημονικού περιεχομένου των ε, κοινών επιτροπών των συμφωνιών ελευτικής σύμπραξης. Έτσι λοιπόν, έχουμε εμείς μερικά μόνο εργαστήρια ψήξης ή συσκευασίας νοπού χταποδιού. Αλλά κατά τα άλλα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυξήθηκαν οι δραστηριότητε μας. Εμείς έχουμε κάποιες ερευνητικές δραστηριότητες επί το επιτοπλίστων είχαμε εξοπλισμό σκαφών με χρήματα που πήραμε από διάφορους δανειστές. Τα χρήματα πήγανε κυρίως πάντως στην έρευνα και στον έλεγχο. Λιγότερα για τον εξοπλισμό. ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, δεν βοηθήθηκε η αλία στη χώρα μας. Ενώ υπάρχουν προγράμματα ανατομέα, δεν χρηματοδοτήθηκαν, δεν χρηματοδοτήθηκαν οι τομείς αυτοί. Υπάρχει πρόβλημα απορρόφησης των κονδυλίων και η κυβέρνηση δεν καταφέρει να θέσει σε εφαρμογή τα προγράμματα αυτά. Τα χρήματα τα χρησιμοποιούμε μερικέ φορέ για κοινωνικά μέτρα που δεν είναι ο καλύτερο τρόπο για να βοηθήσουμε την αλία. Οι πόροι υπάρχουν ανατομέα. Δεν χρησιμοποιούνται όμως καλά, χάνονται. Υπάρχουν ανάγκες που δεν χρηματοδοτούνται. Δεν υπάρχει καλή διαχείριση λοιπόν των κονδυλίων ανατομέα. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι πολλές εκατοντάδες ε, πλοίων δραστηριοποιούνται στα έδατα της Μαυριτανίας περιορίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την εσωτερική αλία. Μαθηματικά είναι αδύνατον όσο αποτελεσματικά και αν είναι τα μέσα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα σκάφη που δραστηριοποιούνται στην αλία μικρής κλίμακας. Είτε πρόκειται για εμπορικά, είτε πρόκειται για τις απορρίψεις κλπ. Τα αποτελέσματα δεν μπορούν παρά να είναι ελάχιστα. Θα έρθω τώρα λιγάκι στην Κίνα Και γιατί. Διότι έχει χρηματοδοτήσει η Κίνα την ανανέωση του στόλου της και αλλιεύει στη ύδατα της Μαυρητανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε ό,τι έπρεπε. Σε επίπεδο τοπικό, ενώ η Κίνα χρηματοδοτεί προγράμματα για 100 εκατομμύρια δολάρια για τη μεταποίηση. Υπάρχει λοιπόν πρόγραμμα για τα μικρά πελαγιακά είδη, το οποίο, πρόγραμμα αυτό της Κίνας επιτρέπει στην Μαυριτανία να ε, εξοπλίσει καλύτερα το στόλο της. Ψυχολογικά είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, τι γίνεται για το μέλλον. θα σας μιλήσω για μια χάρτα χρηστής διακυβέρνησης που προτείνουμε εμείς με την οποία πρέπει να δεσμεύονται όλες οι πλευρές. Η κυβέρνησή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρξει μία δίκαια κατανομή των πόρων. Αν δεν υπάρχει δίκαια κατανομή του πλούτου αυτού, δεν συμφέρει την Μαυριτανία να προχωρήσει σε συμφωνίες αλληλευτικές σύμπραξης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει λίγο περισσότερο την ανάπτυξη του τοπικού πληθυσμού. Να υπάρξει αυτή η προστιθέμενη αξία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, δόκτωρα Μούντ Σερίφ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπρέτ Φίσκνετ, που είναι από την ώρα εμπειρογνώμων. Εμπειρογνώμων στην Αλία τα τελευταία 30 χρόνια και στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα. Περιμένουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει για τις αλλιευτικές συμφωνίες σύμπραξης. Thank ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για το ότι προσκαλήσατε την Νούνταρτ να έρθει εδώ να προσέλθει σε αυτή την ακρόαση και να δώσει μια σύντομη επισκόπηση για την βοήθεια στην ανάπτυξη στον τομέα της αλληλείας από την Νορβηγία. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την πολιτική αλληλείας της Νορβηγίας, όχι για την ανάπτυξη, αλλά συμφέροντος νορβηγικού κατά κάποιο τρόπο. Η Νορβηγία δεν έχει διμερείς συμφωνίες με αναπτυσσόμενες χώρες για να έχει πρόσβαση στους πόρους, στους αλληλευτικούς πόρους. Είναι απόφαση επί της αρχής αυτή η πολιτική απόφαση για να είναι βιώσιμη η αλληλεία, περισσότερο οικονομικά βιώσιμη, θεωρήθηκε αναγκαίο να μειωθεί ο αριθμός των σκαφών που α, αλίευε από πλευράς Νορβηγίας, ευθυγραμμιζόμενη στη μείωση του δυναμικού των ε, αλευτικών στόλων, όπως είχε συμφωνηθεί από την Αρμόδια Επιτροπή το 1999 για την Αλία. Οι διαθωτικές αυτές προσαρμογές λοιπόν όσον αφορά τον στόλο μας για την Αλία το 2005 και το άνοιγμα της μεταφοράς ε, ποσοστώσεων από ένα σκάφος σε άλλο υπό τον όρο ότι θα αφαιρεί το από την ε, αλλιευτική δραστηριότητα ένα σκάφος το οποίο δεν θα είχε πλέον τέτοια ποσόστοση και δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αλλού. Πράγμα το οποίο θα σήμαινε την μεταφορά της υπεραλίευσης με αυτόν τον τρόπο σε, κάποιο, σε κάποια άλλη ζώνη. Επιπρόσθετα, είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι πλοία που έχουν νεολογηθεί στην ε, Νορβηγία δεν επιτρέπεται να αλλιεύουν ε, εκτός υδάτων ε, νορβηγικής αρμοδιότητας, εκτός αν υπάρχει η συμφωνία όπως στην ΝΑΦΟ, Κομελάρ κτλ. Τώρα να στραφώ στην πολιτική για την ανάπτυξη από πλευράς της Νορβηγίας. Η πρώτη υποστήριξη στην ανάπτυξη που δόθηκε από την Νορβηγία ήταν το 1952 στον τομέα της Αλίας στην Ινδία, στην Κεράλα. Και ένα άλλο πρόγραμμα ήταν το πρόγραμμα Nansen, όπου το ε, ερευνητικό σκάφος of Nansen χρησιμοποιήθηκε σε παγκόσμια κλίμακα για να αξιολογηθούν ε, οι αλλιευτικοί πόροι. Και έτσι φτάνουμε στο 1973 σε συνεργασία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και με τον ΦΑΟ. Και από το 2007 συνέχισε υπό την αιγίδα του ΦΑΟ ως ε, το πρόγραμμα του ε, of Νάνσεν, το ε, οικολογικό πρόγραμμα όσον αφορά την αλληλεία με συμμετοχή σε διεθνές πλαίσιο για την οικολογική προσέγγιση όσον αφορά την αλληλεία, την περιβαλλοντική προσέγγιση, υποστηρίζοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες να καταστήσουν λειτουργική αυτή την προσέγγιση στις πολιτικές τους. Επίσης, η επικέντρωση είναι στην έρευνα, στην αξιολόγηση των αποθεμάτων, στην εκπαίδευση και παιδεία όσον αφορά τα αλλιεύματα και στην θεσμική οικοδόμηση ως αναγκαίους όρους για να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική. Στη συνέχεια, επικεντρωθήκαμε περισσότερο <clears throat> στην καταπολέμηση της ε, παράνομης ε, και ε, μη συμβατής αλληλείας, UU αλληλείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και από πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Τώρα, στη συνέχεια, κάποια μεγαλύτερα προγράμματα, εγχειρήματα όσον αφορά την υποστήριξη στην Αλία έδωσαν λόγω κάποιων στρεβλών ή μη ορθών διαδικασιών όχι και τόσο καλό όνομα στην Αλία. Μεγάλες ε, αλία, ε, επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα και όπου από πλευράς της κυβέρνησης ε, η συμμετοχή όπως μπορείτε να ενθυμηθείτε ήταν μεγαλες αλί ιδιαίτερα στον παραγωγικο τομεα και οπου απο πλευρά της κυβερνησης η συμμετοχη τομέα με αναπτυσσόμενες χώρες. Απέτυχαν αυτές οι προσεγγίσεις για διάφορους λόγους. Προφανώς ε, ιδιαίτερη σημασία ήταν η απουσία προβληματισμού για την θεσμική και οικονομική αηφορία αυτών των ε, εγχειρημάτων μετά τη δρομολόγησή τους. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 μετακινηθήκαμε περισσότερο στη θεσμική ε, διάρθρωση και οικοδόμηση και όσον αφορά τις κυβερνήσεις να υποστηριχθούν κυβερνητικοί μηχανισμοί και προσεγγίσεις. Ανεξάρτητη αξιολόγηση όσον αφορά τα τελευταία 20 χρόνια από πράσινη της Νορβηγίας υπευλήθη το 2009 και έδωσε μια πιο θετική εικόνα συνολικά. Η σημερινή κυβέρνηση συνασπισμού που πέρυσι ε, δρομολογήθηκε, είπε ότι είναι προτεραιότητα να, βοηθηθεί, να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, στην ανάπτυξη της προσπάθειας της αλίας ε, και της εποπτείας αλίας ως συνεισφορά κατά της παράνομης και παραβατικής αλίας. Για να αναφερθώ σύντομα σε, κάποιες, σε κάποιες συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης, αυτό που εντοπίστηκε ήταν ότι και θεωρήθηκε γενικά θετικό ήταν ότι η ευθύνη για ένα πρόγραμμα θα είναι της χώρας αυτής, της αναπτυσσόμενης χώρας και θα επικουρεί η Νορβηγία στην υλοποίηση του προγράμματος. Υπάρχει μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση σε ένα χρονοδιάγραμμα 15-20 ετών, σε ένα χρονορίζοντα ευρύτερο η ευθύνη και η ανάγκη ανταπόκρισης όσον αφορά μεταβαλλόμενους όρους και προϋποθέσεις σημαίνει ότι η αναπτυσσόμενη χώρα θα είχε τα ενία στα χέρια της και σε περίπτωση κάποιων μεταβολών το πρόγραμμα αυτό θα προσαρμοζόταν, θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές και να προσαρμόζεται σε αυτές και, μια πιο ανοιχτή σε σχέση με τον ε, προγραμματισμό ε, προσέγγιση και στον προγραμματισμό και σχεδιασμό και στην υλοποίηση. Τα ίδια θεσμικά όργανα ασχολούνται σε σχέση με το σχεδιασμό και με την ε, υλοποίηση των σχεδίων αυτών. Αυτό είναι δυνατόν και είναι εφικτό επειδή χρησιμοποιούμε τα, ε, τις διευθύνσεις ε, και το ε, στελεχειακό δυναμικό των δικών μας Υπουργείων όσον αφορά αυτές τις πρωτοβουλίες. Οι ίδιοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων και στην σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων και στην υλοποίησή τους. Η ενίσχυση των θεσμικών εθνικών οργάνων είναι η κύρια επικέντρωσή μας. Εστιαζόμαστε ιδιαίτερα σε αυτό. Τώρα στη συνέχεια θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία παίρνει διάφορες ε, μορφές ε, πολυσχηδώς και έχουμε εδώ μια παρήθμιση των χωρών με τις οποίες ε, η Νορβηγία έχει διμερή συνεργασία, κάποιες χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής για παράδειγμα. Οι μεγαλύτεροι, οι κυριότερες συνεργαζόμενες χώρες είναι η Μοζαμβίκη, όπου έχουμε ένα πρόγραμμα ειδικό για την Αλία και το Βιετνάμ, όπου είχαμε και μακρόχρονη συνεργασία με αυτή τη χώρα μέχρι σήμερα, περιφερειακά προγράμματα στη συνέχεια. Και όλα αυτά συχνά είναι απόρρια, είναι επίπτωση της συνεργασίας, διμερού συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο. <clears throat> Για την Νοτιοδυτική Αφρική, για παράδειγμα, μεταξύ Αγγόλας, Ναμίβιας και Νότιας Αφρικής, ξεκινώντας ένα τέτοιο πρόγραμμα που ξεκίνησε στις αρχές του 1990 και με τις οποίες χώρες είχε και διμερή συνεργασία. Η Νορβηγία είναι ένα παράδειγμα σχετικά. Μετά, συγγνώμη, έχουμε και δύο άλλα προγράμματα όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές και την ικανότητα για τις τοπικές κοινότητες να μπορούν να προσαρμόζονται σε αυτές τις κλιματικές αλλαγές. Έχουμε επίσης και μια πιο μακρόχρονη σειρά στοιχείων που έχουν συλλεγεί επί 20 χρόνια μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Nansen για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες τάσεις σε αυτές τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και να προσαρμοστεί κανείς σε αυτά τα στοιχεία στις κλιματικές αλλαγές. Και μετά και υποστήριξη όσον αφορά την πολυμερή συνεργασία έχουμε κάποια ε, προγράμματα εκεί και με τον ιδιωτικό τομέα που επίσης ε, υποστηρίζεται με κονδύλια από πλευράς ε, των νορβηγικών οργάνων. Τώρα, η κύρια κατεύθυνση που ακολουθούμε στην συνεργασία για την ανάπτυξη ποια είναι. Είναι να συνεισφέρουμε στην αηφόρο χρήση των πόρων όσον αφορά την φύση και το περιβάλλον. Ουσιώδες είναι εδώ οι αποφάσεις για τη διαχείριση να βασίζονται σε επιστημονικά τεκμήρια, επιστημονικά στοιχεία και αναλύσεις και να είναι να συνάδουν σαφώς με διεθνείς ε, συμβάσεις ε, και διατάξεις ε, και νόμους. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τα θεσμικά όργανα, τα εθνικά, που είναι σημαντικά και για την περιφερική συνεργασία. Οι εμπλεκόμενοι, όσοι ενέχονται, θα πρέπει να εισακούγονται όσον αφορά τις απόψεις τους για τις διάφορες δράσεις και δραστηριότητες και να εστιαζόμαστε στη διαφάνεια και στην χρηστή διακυβέρνηση και χρηστή διαχείριση. Η περιφερειακή υποστήριξη προς, ε, για την ανάπτυξη είναι μια προσέγγιση όπου θα προσεγγίσουν οι χώρες αυτές ε, την ε, Νορβηγία ώστε να τη συνδράμει παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη για την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων. Και τώρα στη συνέχεια θα ήθελα να σας δείξω μια συνολική εικόνα χαρτογράφησης του προγράμματος Νάνσεν που για πολλές χώρες είναι η μόνη πληροφορία που είναι διαθέσιμη για αυτές από πολλές πηγές. Είναι, δείχνει που ήταν, ποια σημεία ήταν κέντρα βάρους τα τελευταία χρόνια η φάση της θεσμικής ε, οικοδόμησης και εδώ έχουμε το πρόγραμμα Νάνσεν για τη συνεργασία με διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο, στο σύστημα της ε, διασφάλισης οικοσυστημάτων και βιοτόπων. Προκλήσεις. Θεωρούμε ότι οι κυριότερες προκλήσεις εδώ και το σημαντικότερο στοιχείο είναι η πολιτική βούληση και το δυναμικό φυσικά δραστηριοποίησης για να ε, ρυθμίσουμε το θέμα των πόρων. Φυσικά οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι και πρέπει να βρούμε τον πιο αποτελεσματικό βέλτιστο τρόπο για την πιο αποτελεσματική διαχείρισή τους και εκμετάλλευσή τους. Περιφερειακή συνεργασία είναι κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να διαχέονται πληροφορίες και να τις μοιράζονται οι εμπλεκόμενοι και μετά να εφαρμόζονται οι διατάξεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις τώρα. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Αλίας και μετά από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ο κύριος Παλέσσα έχει το λόγο. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, porozumienia o rybołówstwie z krajami trzecimi, w szczególności w segmencie οι συμφωνίε για την Αλία με τρίτε χώρε όσον αφορά την, τον κοινοτικό στόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουμε λόγο για το Μαρόκο και τη Μαυριτανία, αυτέ οι συμφωνίε με αυτέ τι χώρε έχουν μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα ιδιαίτερη σημασία για το στόλο αυτό και για τις επιχειρήσεις και για τις αναπτυσσόμενες βέβαια χώρες και στην Δυτική Αφρική. Σε αυτές τις συμφωνίες λοιπόν που είναι καλές για την μία πλευρά και για την άλλη, για αμφότερες τις πλευρές και θέλω εδώ να τονίσουμε και το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν έρχεται η ώρα της εφαρμογής αυτών των ε, συμφωνιών, βλέπουμε κάποια θέματα τα οποία δημιουργούν προσκόμματα ή εμπόδια. Για παράδειγμα, όσον αφορά την μη τήρηση κάποιων διαδικασιών ή όσον αφορά το θέμα της διαφάνειας, πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Με τη Μαυριτανία στην τελευταία μεικτή επιτροπή αντιμετωπίσαμε προβλήματα όπως την έλλειψη διαφάνειας ε, που αφορούσε για παράδειγμα τους ελέγχους ε, των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υλοποιούνται αυτές ε, οι, αυτοί ή το boarding, τα boardings όπως λέγονται στα αγγλικά, οι, οι επί τους ε, έλεγχοι με την παρουσία αξιωματούχων ή και με την εμπλοκή των εφοπλιστών σε αυτούς τους ελέγχους. Και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε ήταν η απουσία, η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το κέντρο εποπτείας ε, επιτήρησης της ε, Μαυριτανίας ε, υλοποιώντας αυτούς τους ελέγχους. Αυτά έχουν τεράστιες επιπτώσεις όμως για τους εφοπλιστές, διότι τους λέγεται ότι σε σχέση με τους αναγκαίους ελέγχους ε, που ε, ε, δεν μπορούν να διεξαχθούν ή για τις κλειστές ζώνες όπου δεν μπορούν να αλλιεύουν. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς υλοποιείται, πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα, πώς μπορεί να υπάρξει μια ε, εγγύηση, να υπάρξουν εχέγγυα, ώστε η, ο στόλος της κοινότητας στα ύδατα της Μαυριτανίας να μπορεί απρόσκοπτα να αλλιεύει. Τι θα κάνει δηλαδή η Μαυριτανία για να, να σεβαστεί τις διατάξεις αυτού του πρωτοκόλου. Όσον αφορά την συμφωνία με το Μαρόκο, θα ήθελα να πω σε σχέση με τι σημερινέ τις και τις μελλοντικέ συμφωνίες, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κάποιο τις προτιμήσεις ε, σε σχέση, θα υπάρξει κάποια προτίμηση εκείνους τους στόλους της Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιούν όλες τις διατάξεις των πρωτοκόλων και τι θα γίνει με το 5% και άλλα σημαντικά θέματα από πλευρά ρητρών για τον κοινοτικό στόλο. Ευχαριστώ. I should like to ask Madame Fisknes. Fisknes. Γνωρίζετε πόσο η νορβηγική πολιτική βοήθεια των αναπτυσσομένων χωρών να αναπτύξουν τον ελευθερικό του κλάδο, πόσο κοστίζει ετησίω και για πόσε χώρε έχετε στοιχεία. Συνέχεια κυρία παρακαλώ. Συγγνώμη, συγγνώμη, κάποια παρανόηση υπήρξε. Λοιπόν, πολύ καλά. Έχω μια ερώτηση προς ε, τον κύριο Μουριέλ, αλλά και ερώτηση προς τον κύριο Σαρίφ. Ξεκινώ με τον κύριο Μουριέλ. Είπατε πιο πριν ότι η συμφωνία, οι συμφωνίες πρέπει να ε, αναδιατυπωθούν ή να εξειδικευτούν. Μπορείτε να τα συγκεκριμενοποιήσετε αυτά τα σχόλιά σας. Ποιες συμφωνίες εννοούσατε. Είπατε ότι το στόλο από 200 σε 100 σκάφη τον περιορίσατε το στόλο. 50% μείωση. Θα μπορούσα να πω αυθόρμητα συγχαρητήρια κύριε. Τι γίνεται όμως με τον όγκο των αλλιευμάτων. Μειώθηκε ο όγκος αλλιευμάτων κατά 50% κατά το ίμιση ή μήπως διπλασιάστηκαν τα αλλιεύματα. Ποιοι κανόνες ελέγχων υφίστανται όσον αφορά την αλληλεία της αλλιευτικές δραστηριότητες σε τρίτες χώρες. Μπορεί να φανταστεί κανείς ότι η ε, βιομηχανία μεταποίησης ή ε, η βιομηχανια αλληλείας ε, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε τέτοια ερευνητικά μέτρα ή ε, τέτοιες δράσεις. Ο κύριος Σαρίφη είπε ότι δεν ε, λειτουργούν εταιρικά αυτές οι συμφωνίες σήμερα. Ερώτησή μου προς εμάς κύριε Μουριέλ, τι προσφέρετε στους εμπλεκόμενους ώστε να διασφαλιστεί μια εταιρική σχέση και συνεργασία με αυτούς. Προς τον κύριο Σαρίφ στη συνέχεια έχω τις εξής ερωτήσεις. Κατά πόσο έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις εταιρικών συμφωνιών σε ανταγωνισμό όμως με άλλες χώρες που αλλιεύουν σε αυτά τα ύδατα με αντίστοιχα δικά του συμφέροντα. Δεύτερη ερώτηση. Ποιε βελτιώσει προβλέπετε και μπορούν να γίνουν στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, όπω βλέπετε και θεωρείτε εσεί, ώστε τα χρήματα που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο πριν ακούσαμε το εντυπωσιακό ποσό 150 λέει ο Μιλήτρια για τα 160 εκατομμύρια να χρησιμοποιούνται σωστά αυτά τα χρήματα και πώ μπορούν αυτά η χρήση του να ελέγχεται πιο αποτελεσματικά. Και τελευταία μου ερώτηση, σε πολλές χώρες του τρίτου κόσμου δεν υπάρχουν δημοκρατικές υποδομές. Ε, τι μπορεί να γίνει ώστε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς εννοούμε, να μπορέσει να, βασίζεται, να βασιζόμαστε εμείς στην υλοποίηση αυτών των ε, συμφωνιών. Υπάρχουν κάποια μέσα, όπως βλέπετε εσείς, που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιτευχθεί ο στόχος. Ευχαριστώ. Κύριε το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα στον κύριο Σερίφ επίσης. Μιλούσατε, λέγατε ότι η Μαυριτανία δεν έχει την ικανότητα να ελέγχει τι κάνουν τα αλλιευτικά πλοία κτλ. Ε, το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται, ώστε να ξέρουμε για τι δυναμικό μιλάμε και επίση ε, πω γίνεται συνεργασία με τους τόλου, Σας δίνουν δηλαδή τι απαραίτητε πληροφορίες, σας αφήνουν εν πλώ, αν θέλετε να ελέγξετε το πλοίο κτλ. Και επίσης μπορείτε να μου πείτε και οι άλλοι στου ομιλητέ, μιλάμε για την αναμόρφωση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Τι θέλετε εσείς, τι επιθυμείτε, τι προτείνετε εσείς από τη δική σας σκοπιά, τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά αφού επισημάνατε τα προβλήματα, ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Επισημάνατε προβλήματα. Τι πιστεύετε θα μπορούσαμε να κάνουμε ή τι μπορούμε να κάνουμε. Από πλευρά Νορβηγίας είπατε ότι ορισμένα πράγματα γίνονται καλά στην Νορβηγία, αλλά τι θα μας συνιστούσατε να πάρουμε από τη δική σας την εμπειρία εμείς. Ευχαριστώ. Η Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ, έχουν γίνει διάφορες ερωτήσεις, θα ήθελα να διατυπώσω την πρώτη προς την κυρία Ζολή. Έγινε μια εισαγωγή υπό το πρίσμα της Επιτροπής Ανάπτυξης από πλευρά της. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική της Επιτροπής Ανάπτυξης αυτή η προσέγγιση. Είναι σημαντικό νομίζω να το ταυτοποιήσουμε αυτό και να το εντοπίσουμε με ένα σημαντικό φορτίο πολιτικής, ή πολιτικό φορτίο όσον αφορά τις συμφωνίες αλληλείας. Κάνουμε λόγο για την εξωτερική διάσταση της κοινή ε, αλληλευτικής πολιτικής και στην Επιτροπή Αλίας. Και νομίζω ότι και οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, εμείς εδώ στην Ευρωβουλή θα έπρεπε να ενώσουμε τα δύο αυτά κριτήρια της ευθύνης, της υπευθυνότητας και της αηφορίας. Στις συμφωνίες αλίας έχουμε δύο τμήματα. Εσείς πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Είναι η καθαρά εμπορική συμφωνία και η βοήθεια προς την ανάπτυξη αυτό το τμήμα της βοήθειας προς την ανάπτυξη. Οι συμφωνίες οι σε ένα τμήμα τους καθαρά αναφέρονται σε ένα άρθρο των Ηνωμένων Εθνών στο οποίο γίνεται αλληλεία όσον αφορά τα πλεονάσματα. Σήμερα το πρωί έγινε μια παρέμβαση και αναφέρεται αυτό εφόσον δεν θα υπάρχει και καμία στρέβλωση στη ζώνη εκείνη όπου θα ασκείται η ελευτική δραστηριότητα και με κριτήρια αντιστάθμισης. Εδώ λοιπόν θα πρέπει πάλι να αξιολογήσουμε τη βοήθεια προς την ανάπτυξη, πώς γίνεται και με ποιο τρόπο διαμορφώνεται. Δεν πιστεύω ότι η μία επιτροπή μπορεί να διαμφισβητεί την άλλη. Είναι σημαντικό να διαφοροποιούμε αυτά τα δύο θέματα και πρέπει με μια αρχή συνεκτικότητας ε, και ε, συνοχής να μπορούμε να δρούμε. Διότι εδώ γίνεται λόγος για χώρες, για παράδειγμα όπως ε, για την Ισπανία. Έχουν αμφισβητηθεί τα θέματα, για παράδειγμα, επιστημονικών τεκμηρίων. Θα ήθελα να ξέρουμε τι γίνεται εδώ σε σχέση με την μία αρχή, το ένα σώμα ή το άλλο Πρέπει να υπάρχει όμως μια, ένα κριτήριο συνοχής και συνεκτικότητας μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτοπών μας. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Στον επόμενο γύρο των παρεμβάσεων θα ήθελα να διατυπώσω κάποια άλλη ερώτηση στους εισηγητές. Ευχαριστώ. I, I think that this... Νομίζω ότι η συνάντηση αυτή ήταν πολύ σημαντική γιατί συνειδητοποιούμε σε τι κρίση βρισκόμαστε. Συνειδητοποιούμε, ακούσαμε από τους εμπειρογνώμονες τι γίνεται με τα αποθέματα, αλλά και εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι το μείγμα που έχουμε, αλλιευτικές συμφωνίες, που προσπαθούν να είναι και συμφωνίες αναπτυξιακές, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών μελών της Επιτροπής Ανάπτυξης, δεν είναι ότι καλύτερο. Πρέπει να χωριστούν αυτές οι δύο πτυχές των συμφωνιών και να έχουμε οι καθαρά αναπτυξιακές συμφωνίες, οι ελευτικές συμφωνίες, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ένδια αν προσπαθούμε να τις συνδυάσουμε τις αναπτυξιακές συμφωνίες με την πρόσβαση στους πόρους, αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Γιατί δείχνει ότι τελικά έχουμε άλλες βλέψεις. Λέμε ότι το κάνουμε για την ανάπτυξη, αλλά τελικά δεν είναι για την ανάπτυξη. Η πρώτη τέτοια συμφωνία που είδε ήταν εκείνη με την Κινέα, όπου είμαστε έτοιμοι να δώσουμε χρήματα στους ανθρώπους εκεί. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να το καταλάβουμε αυτό. Και είναι σοβαρό. Αυτό που πρέπει τώρα να στοχεύσουμε είναι να έχουμε μια υφόρο αλία, να έχουμε χρηστή διακυβέρνηση και να καταπολεμήσουμε την ένδια. Δεν είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τι έχει γίνει στη Δυτική Αφρική, ότι δεν ήταν ανάπτυξη. Ήρθε λοιπόν η στιγμή για μια νέα αλλιευτική πολιτική που θα έχει αναπτυξιακές συμφωνίες χώρια από τις αλλιευτικές. Δεν μπορεί να λέμε ότι κάνουμε ανάπτυξη στην Κινέα όταν προσπαθούμε να δώσουμε 300.000 στους ανθρώπους που σκότωσαν 172 ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρά αυτά. Σίγουρα είναι και πολιτικά φορτισμένη οι αποφάσεις μας, αλλά να ξέρουμε ότι άλλο η ανάπτυξη, άλλο η αλεία. Η αλεία είναι ένα πολύ σημαντικό σκέλος της ανάπτυξης, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε την αηφόρο αλεία επιστημονικά, ώστε να λάβουμε υπόψη μας όσα λένε οι επιστήμονες και όχι να συνεχίσουμε να τα κάνουμε τα πράγματα όπως τα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Αν δείτε τι απέδωσε η αλληλευτική μας συμφωνία με την Κινέα είναι τρομερό. Δεν μπορείτε να κλείνετε τα μάτια σε μια τέτοια πραγματικότητα και αλήθεια. Η κυρία Λοβίνη έχει τώρα το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Επειδή, κυρίες Πρόεδρε, επειδή ανήκω στις δύο επιτροπές. Λοιπόν, πράγματι. Εδώ όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μίλησαν που παρουσίασαν μια ευρία εικόνα ε, και όλες τις πλευρές του θέματος. Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την αναμόρφωση της κοινή ελευθερικής πολιτικής όσον αφορά το εξωτερικό της σκέλος. Εάν δούμε την σημερινή εξωτερική πολιτική ε, στα πλαίσια των συμπράξεων, αν θέλετε, ποιοι είναι οι στόχοι. Οι στόχοι είναι τρεις που διατυπώθηκαν. Πρώτον, να υπάρξουν ε, αλληλευτικές ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό στόλο. Δεύτερον, να παράσχουμε αλία στην ευρωπαϊκή αγορά και τρίτον, να προωθήσουμε την αηφόρο αλία στις συμβαλόμενες χώρες. Αυτοί οι τρεις στόχοι, ή τουλάχιστον δύο από τους τρεις, μπορούν να συζητηθούν. Οι δύο πρώτοι στόχοι. Δηλαδή να δημιουργηθούν αλληλευτικές ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό στόλο, πληρώνοντας για πρόσβαση ε, στα αλληλευτικά ύδατα από μέρους των φορολογουμένων και των 27 κρατών μελών, ενώ γνωρίζουμε τα δύο τρίτα των συμφωνιών πρόσβασης χρησιμοποιούνται από μία χώρα, την Ισπανία. Και από τη χώρα μου, η χώρα μου τουλάχιστον δεν χρησιμοποιεί όλες τις συμφωνίες. Λοιπόν, μας είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στον ε, Σουηδό φορολογούμενο ότι θα πρέπει να πληρώνει για αυτή την πρόσβαση. Με χαρά άκουσα από τον κλάδο ότι είναι λογικό ότι και ο κλάδος θα πρέπει να πληρώσει για την πρόσβαση. Ως εδώ εντάξει. Αλλά τώρα, η προμήθεια της ευρωπαϊκής αγοράς με ψάρια. Ε, ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από αυτές τις συμφωνίες και ήδη η Επιτροπή ανέφερε ότι αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή αυτής της αλίας και δεν χρειάζεται ε, οι Ευρωπαίοι αλλοί να ψαρέψουν. Μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή ψαριών από τις τρίτες χώρες και να κάνουμε και οικονομίες. Δεν νομίζω ότι από οικονομική άποψη ευσταθεί αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν, να προωθήσουμε μία αηφόρο αλία στις συμβαλόμενες χώρες. Ναι, ναι, εδώ συμφωνώ. Όλοι οι φορολογούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμφωνήσουν. Ε, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος των συμφωνιών μας. Συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Γκόρες ότι πρέπει να υπάρξει χρηστή διακυβέρνηση, μια συμφωνία πλαίσιο περί χρηστή διακυβέρνηση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει στην έρευνα, στον έλεγχο και στην πρόθεση της αλίας στις χώρες του τρίτου κόσμου ή στις παράκτης χώρες. ανεξάρτητα από το αν υπάρχει πρόσβαση ε, στην αλία από τα ε, ευρωπαϊκά πλοία. Σε αυτά τα είδατα δηλαδή. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα και με την Νορβηγία η οποία δεν το ανέφερε αλλά ε, χρηματοδοτεί το μόνο πλοίο το οποίο κάνει επιστημονικές έρευνες και εκτιμήσεις των αποθεμάτων στα είδατα της Δυτικής Αφρικής. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μπορείτε να μου απαντήσετε στο ερώτημα και σας το θέτω, κυρία Σίκνες, αν νομίζετε ότι οι εκτιμήσεις αποθεμάτων ε, στα, στις ακτές της ε, Βόρειας Αφρικής αρκούν για να δούμε κατά πόσον υπάρχει πλεόνασμα ηχθείων που μπορούν να πουλήσουν αυτές οι χώρες στα πλαίσια των ελευθερικών συμφωνιών. Διότι αυτό συμφωνεί με το δίκαιο της θάλασσας του ΟΗΕ. Δηλαδή ότι οποιαδήποτε χώρα μπορεί να πουλήσει φυσικά ε, τους αλληλευτικούς σπόρους εάν υπάρχει πλεόνασμα Αλλιώς και ο τοπικός πληθυσμός αυτής της χώρας δεν χρειάζεται να καταναλώσει αυτό το ψάρι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν συνάπτουμε τις συμφωνίες. Να μπορούμε να θεσπίσουμε ότι θα υπάρχει ένα πλεόνασμα και τι θα γίνει με το πλεόνασμα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει τα, τα χρήματα υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιούνται σωστά για επιστημονική έρευνα, όπως είπαμε, και για τον έλεγχο. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα ε, στη Δυτική Αφρική. Αυτά, αυτή είναι η πρώτη μου αντίδραση. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. Τώρα θα ήθελα να κάνω και ορισμένε ερωτήσεις. Στρέφομαι στην Επιτροπή. Επειδή προσπαθώ να βρω ως προς τη διαφάνεια, ποια είναι η συνολική αξία των ε, συνολικών συμπράξεων. Ποια είναι η τιμή, η αξία, η αξία of the fish that comes from these agreements. Των εκφορτώσεων, ποια είναι η αξία, δηλαδή σε ποιες χώρες πηγαίνουν, στην Ευρώπη, Και στον κύριο Σερίφ από τη Μαυριτανία θα ήθελα ρωτήσω το εξή. Γνωρίζουμε ότι ο 1 τρίτο του κρατικού προπολογισμού στη Μαυριτανία προέρχεται από τι Ευρωπαϊκέ Αλληλευτικέ Συμφωνίε. Έχω επισκεφθεί τη Μαυριτανία πριν από λίγο καιρό και γνωρίζοντα ότι το 50% αυτού του 1 τρίτου έχει ως αντικείμενο να υποστηρίξει την τοπική αλία και τη διαχείριση και την πρόθεση της αλίας στη Μαυριτανία οι αλήσει του οποίους είδα δεν είχαν ε, σωσίβια, δεν ε, γνώριζαν τα λιμάνια ε, στις ακτές Μαυριτανίας και μάλιστα έχουν κίνδυνο να πνιγούν και πολλοί πνίγονται, συνεχώς θα έλεγα πνίγονται. Οι περισσότεροι είναι αναλφάβητοι και δεν ε, ήξεραν πώς να κάνουν πρόγνωση καιρού ή να ζητήσουν την πρόγνωση του καιρού. Ε, προσπάθησα λοιπόν να δω ε, τι γίνεται, εάν έχω ένα σύστημα προϋποειδοποιήσεις για κακοκαιρία στις ακτές, αλλά ε, τα πλοιάρια τους ήταν πολύ πρωτόγωνα. Λοιπόν, κύριε Σαρίφη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθύνονται προς την πρόθεση ε, της αλίας και των αλλιέων στη Μαυρετανία. Πιστεύετε ότι ε, όταν υπάρχει μεικτή αλία ή μεικτά είδη μαζί με τα ευρωπαϊκά πλοία ανταγωνίζονται τους τοπικούς αλίες ή παίρνουν, παίρνουν δηλαδή κάτι το οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι οι τοπικοί αλίες. I think the floor is for Madame Keller. Κυρία Κέλλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δευτερολογώ, αλλά ορισμένοι συνάδελφοι ή πολλοί αναφέρθηκαν ε, στην ανάγκη συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών. Και ε, στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας έχουμε νέες ευθύνες, αλλά και έχουμε και περισσότερες υποχρεώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν όλα υπόψη όταν γίνεται αναμόρφωση της ε, αλληλευτικής πολιτικής. Και ευτυχώς η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται ε, στην υποχρέωση για συνοχή και λέει ότι καμία πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να είναι αντίθετη προς τους αναπτυξιακού στόχου και ο πρώτος είναι η εξάλληψη τη φτώχεια. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πούν οι ομιλητές ε, κατά πόσο πιστεύουν ότι αυτή η κοινή αντιευτική πολιτική που μας απασχολεί είναι συνεκτική με την ανάπτυξη. Όταν λέω συνεκτική, όχι με την ανάπτυξη, αλλά αν βοηθάει την ανάπτυξη. Δηλαδή, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι. Gracias, Presidenta. Ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ να στηρίξω ξεκάθαρα τον ευρωπαϊκό αλληλευτικό τομέα. Νομίζω ότι έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του ευρωπαϊκού κλάδου. που συμμετέχει στις διάφορες διεθνείς συμβάσεις. Από όσο ξέρω, λοιπόν, πρέπει να στηρίξουμε τον κλάδο που συμπεριφέρεται υπεύθυνα και που θέλει να συνεχίσει να ζει από τη θάλασσα. Άρα Πρέπει να υπάρχουν οι καλύτεροι δυνατόν έλεγχοι για να αποφύγουμε την παράνομη αλία και τις καλύτερες δυνατόν συμβάσεις με τρίτες χώρες, ώστε κάθε συμφωνία ανάπτυξης να φροντίζει και για την αλία. Επίσης, το Κοινοβούλιο πρέπει να φροντίσει για αυτές τις συμφωνίες, τις αλληλευτικές με τρίτες χώρες να συνεχιστούν γιατί είναι συμφωνίες από τις οποίες ωφέλη έχουν και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι τρίτες χώρες. Επίσης, ο κλάδος αυτός είναι υπέρ και παίρνει ό,τι μέτρα μπορεί ώστε να έχουμε αηφόρο αλία. Δεν θέλει τίποτα περισσότερο από το να κοιτάξουμε τι μέσα χρησιμοποιούν για την αλία, ποιες μεθόδους αλληλευτικές χρησιμοποιούν. Είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια και συμφωνώ με τους ο ομιλητέ μας εδώ στο εξή θέμα. Και μάλιστα θα το ζήταγα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα των ε, συμφωνιών από την αρχή μέχρι το τέλος. Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να γνωρίζουμε ποια είναι τα αποτελέσματα για κάθε χώρα όσον αφορά την ανάπτυξή της. Οι συμφωνίες αυτές δηλαδή σε τι βαθμό βοήθησαν την ανάπτυξή της. Γιατί από αυτά έχει να υποφοληθεί η Ευρώπη, ο αλληλευτικός τομέας, ο οποίος πλήττεται συνεχώς. Πιστεύω λοιπόν ότι η διαφάνεια είναι κάτι από το οποίο έχει να ωφεληθεί και η κοινή αναπτυξιακή μας πολιτική. Θέλω να υπογραμμίσω κάτι από τη σημερινή συζήτηση. Άκουσα την εκπρόσωπο της Νορβηγίας να μας μιλάει για τις εξελίξεις και ναι, καλό, φυσικά και πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις, να στηρίζονται οι τρίτες χώρες, αφρικανικές χώρες, αναφέρθηκε στη συνεργασία με αυτές και τη Μαυριτανία συγκεκριμένα. Συγχρόνως, ο κύριος Αμέτ μας έλεγε ότι επειδή δεν υπάρχουν συμφωνίες με την Ευρώπη ή τόσο πάντων επειδή έχουν μειωθεί, έκανα συμφωνία με την Κίνα και πάει η αγορά. Να λοιπόν η μεγάλη αντίφαση. Ρωτάω λοιπόν την εκπρόσωπο της Νορβηγίας, με αυτή τη στήριξη στην ανάπτυξη, πώς θα ελέγξουμε χώρες της Αφρικής να μην καλύπτουν το κενό που αφήνουμε εμείς από, με άλλες χώρες. Δεν φταίμε εμείς που δεν έχουμε τέτοιες συμφωνίες. Όταν έχουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες, ίσως μπορούμε, αν μη τι άλλο, να επηρεάσουμε τις τρίτες αυτές χώρες και στην ε, Νοτιδυτική Αφρική, ώστε να αποφεύγεται η παράνομη αλία, ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, για παράδειγμα, και οι κανόνες που θα ισχύουν εκεί είναι αυτοί που ισχύουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτά που άκουσα λοιπόν, όχι μόνο σήμερα, αλλά από όλε τι συναντήσει που είχαμε για τη μεταρρύθμιση τη ε, κοινή ελευθερική πολιτική, κατάλαβα ότι ο κλάδο τι ζητάει, ζητάει έλεγχο. Ναι, τρίτε χώρε. Το θέμα είναι να υπάρχει έλεγχος, γιατί σήμερα δεν υπάρχει ο έλεγχος που θα έπρεπε να υπάρχει. Τι θα γίνει, έχουμε αυτές τις καινούριε χώρες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλίας, οι οποίες δεν ελέγχονται. Κάτω από τι προδιαγραφές αλλιεύουν. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει, να δουλέψει, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Γιατί όλοι έχουμε να ωφεληθούμε από τη διαφάνεια. Και η εικόνα του κλάδου της αλίας βελτιώνεται, που δυστυχώς συχνά είναι πολύ αρνητική, και από την άλλη μεριά οι χώρες που εμείς εγκαταλείψαμε δεν θα χρειάζεται να προσφεύγουν σε άλλες χώρες που δεν τηρούν τους κανόνες. Και τέλος, δεν έχω ακούσει ποτέ να μιλάμε τόσο άσχημα για την παγκοσμιοποίηση, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς, ενώ μιλάμε πολύ άσχημα για τον ελευτικό κλάδο συχνά. Όλες αυτές οι σκέψεις πρέπει να συζητηθούν ώστε να έχουμε λογικές αποφάσεις στο μέλλον για μια αηφόρο αλία, για μια αηφόρο οικονομία υπέρ και των τρίτων χωρών, μέσω συνεργασίας μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον όλων, προστατεύοντας όμως και την Ευρωπαϊκή Αλία. Διότι ανάλογα και με, αν συνεχίσουμε με το ρυθμό που πάμε και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σήμερα και την Ελία, αυτή θα εξαφανιστεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ε, κυρία Αντρέα, ναι, αλλά σύντομα παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Έχουμε ή δεν έχουμε αλληλευτικές συμφωνίες. Αν πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίες οι αλληλευτικές συμφωνίες, και για την αναπτυξιακή βοήθεια στις χώρες που υποφέρουν από έλλειψη ανάπτυξης. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να αναλάβει ένα κόστος και η επιχείρηση που δραστηριοποιείται εκεί. Μήπως πρέπει να υπάρχουν κανόνες για πλήρωμα από την περιοχή, για επενδύσεις στην περιοχή και τότε τι διαφορά έχει μια αλληλευτική συμφωνία από μια αλλιευτική αναπτυξιακή συμφωνία που μας ανέφερε η εκπρόσωπο της Νορβηγίας. Εγώ δεν βλέπω ότι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα. Λέμε ότι η αλία είναι εμπορική ευκαιρία και από την άλλη μεριά έχουμε την ανάπτυξη ή αυτά συνδυάζονται. Πρόεδρος, και εγώ έχω κάποια σχόλια και κάποιες ερωτήσεις. Πιστεύω ότι η πολιτική αλληλευτικών συμφωνιών σύμπραξης έχει να κάνει με την αναπτυξιακή πολιτική. Μόνο που ο κύριος στόχος είναι η εμπορική συμφωνία. Βέβαια που συνάδει με την ανάπτυξη. Κατόπιν τούτου, πρέπει να σας πω ότι εδώ μιλάμε για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχουν χώρες μέλη που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ελευτικού τομέα των τρίτων χωρών. Για παράδειγμα, η Ισπανία, μια που αναφέρθηκε, και εγώ θα μιλήσω για την Ισπανία που την ξέρω καλά, γίνεται αξιολόγηση των αποθεμάτων σε τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα στο Μαρόκο, από ισπανικό σκάφος. Εδώ δεν είπαμε τι κάνει για παράδειγμα η Γερμανία στην Αγγόλα ή τι κάνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες Μιλάμε για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκπρόσωπος της Νορβηγίας μίλησε για αυτά που ξέρει από την Νορβηγία. Αλλά πρέπει να προσθέσουμε κάθε φορά τι κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες για να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των τρίτων χωρών μέσω του εθνικού τους προπολογισμού. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει την πρωτοβουλία Πέσκα, που είναι υπέρ της ανάπτυξης και που είναι πολύ περισσότερα από τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα οποία πληρώνονται και οικονομικά ανταλλάγματα. Εμεί μιλάμε εδώ για το κοινοτικό επίπεδο. Αν θέλετε να μιλήσουμε και για τα κράτη-μέλη και τι κάνει το κάθε κράτο μέλο υπέρ τη ανάπτυξη των τρίτων χωρών, να το πούμε. Προ την κυρία Γκόρε τώρα. Για την αηφόρο ανάπτυξη. Εννοείται ότι συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν ευνοϊκέ προποθέσει. Βεβαίω, όλα αυτά συμφωνούμε. Αλλά τελικά είναι η τρίτη χώρα εκείνη η οποία έχει την ευθύνη τη διαχείριση. Εδώ δεν μιλάμε για πικιοκρατία, δεν θα πούμε εμείς τι πρέπει να κάνει μια τρίτη χώρα. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να υπάρξουν οι προποθέσει Να και ο κύριος Βαλέσσα τα είπε πριν. Οι χώρες κάνουν διάφορα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο έχει εγκριθεί και μετά μια τρίτη χώρα λένε ότι η, μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια τρίτη χώρα πάει με διπλό μερίδιο στην αλίευση. Εμείς μιλάμε για την αλίευση από μακριά και έχουμε μια επιστολή που λέει ότι το πρωτόκολλο UBMS δεν είναι αξιόπιστο και ότι υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι ελέγχου. Μα όσοι γνωρίζουν λίγο πολύ τα πράγματα, ξέρουν πολύ καλά ότι όντως υπάρχουν. Για να σας πω ότι μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο, όσο και αν θέλουμε, να επιβάλλουμε προϋποθέσεις υπέρ μιας ε, καλύτερης διαχείρισης των ελιευτικών πόρων. Τώρα, κάτι άλλο που το είπαμε λίγο και σήμερα το πρωί, αλλά επειδή δεν είχαμε κάποιον για την Γρυλανδία, δεν το συζητήσαμε, αλλά θα σας πω τι ρωτήσαμε σήμερα το πρωί και δεν πήραμε απόφαση. Είπαμε, ε, απάντηση. Είπαμε λοιπόν για την Γρυλανδία ότι οι συμφωνίες οι λεγόμενες του Νότου αυτόματα όταν ένα κράτος μέλος δεν χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που του παραχωρούνται αυτόματα αν θέλει κάποιο άλλο κράτος μέλος να ζητήσει τα δικαιώματα αυτά μπορεί να τα πάρει. Αυτό γίνεται με την Γρυλανδία. Θέλω λοιπόν να ξέρω με την ανανέωση των συμφωνιών θα ληφθεί υπόψη αυτό το μέτρο. Η έκθεση αξιολόγησης του 2007 για τις αλληλευτικές δυνατότητες ήταν 58% και 65% 2008. Τι θα γίνει επίση με τη χρηματοδότηση. Μια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι στο μέλλον το εμπορικό τμήμα θα αυξηθεί όσον αφορά τη συμμετοχή των ε, εφοπλιστών. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο και πώς. Θα εφαρμοστεί παντού. Στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω κάτι και τον κύριο Μουριέλ που αναφέρθηκε στην ρήτρα αποκλειστικότητας. Είπε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Τι εννοούσατε κύριε Μουριέλ? Επειδή ήταν σε σχέση με την ρήτρα αποκλειστικότητας. Τέλος, μία ερώτηση που έχει να κάνει με τη διαχείριση των πόρων. Προς τον κύριο Αχμέτ Μάβετ Σερίφ. Κατάλαβα εγώ ότι στη Μαυριτανία ο νόμος ληφτικός, στο άρθρο του 8 υποχρεώνει να έχουν άδεια όλα τα σκάφη που βγαίνουν να λιεύσουν. Της Μαυριτανίας προφανώς. Έχω διαβάσει όμως επίσης, και δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, ότι η άδεια αυτή που δίνεται στα ληφτικά σκάφη της Μαυριτανίας δεν περιορίζει δεν λέει τι θα αλλιεύσουν. Συνήθως όταν δίνουμε μια άδεια λέμε ότι δίνεται η άδεια για την εξή αλία. Στην περίπτωση της Μαυριτανίας από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Οι άδειε δίνονται λευκό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη διαχείριση των πόρων όπως καταλαβαίνετε γιατί αν υπάρχει η λευκή επιταγή, ψαρεύετε ό,τι θέλετε, δεν θα ήταν καλό αυτό για την προστασία των πόρων Μια που έχουμε κάποιον από τον κλάδο εκεί της Μαυριτανής, καλό θα ήταν να μας εξηγήσετε αν όντω έτσι είναι τα πράγματα. Κυρία Τζόλι, μπορούμε τώρα να δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια, για να μας απαντήσουν στις ερωτήσεις και τα σχόλια που ακούστηκαν εδώ. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μουριέλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από το τέλος για την ρήτρα αποκλειστικότητας. Όπως είπα και πριν, εμείς δεν έχουμε δει να συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα πρόσβαση σε πόρους στα πλαίσια ορισμένων συμφωνιών με τρίτες χώρες, γιατί δεν είχε ζητηθεί ο συγκεκριμένος τρόπος στη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλάζουν όμως τα πράγματα. Και τώρα ναι, ζητάμε να έχουμε πρόσβαση στη μια ή την άλλη χώρα. Η ρήτρα αυτή αποκλειστικότητα σημαίνει ότι ανοίγει η δυνατότητα αυτή πρόσβασης εφόσον το ζητάει η τρίτη πρόσβαση εφοσον Όμως, εδώ χρειάζεται λίγο κοινή λογική. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν με το χρόνο. Κάθε φορά που βλέπουμε ότι κάτι δεν είναι καλά σε μια συμφωνία μπορούμε να το αλλάξουμε. Και αυτό ζητάμε εμείς. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τίποτα άλλο. Έπειτα, ακούσαμε ότι υπάρχουν χώρες που συνεργάζονται στην μελέτη των πόρων. Το επιθυμήσατε κι εσείς κύριε Πρόεδρε ότι η Ισπανία έχει ένα σκάφος το οποίο κάνει τέτοιες έρευνες. Ήταν σε Σενεγάλη μάλιστα πρόσφατα. Το σκάφος αυτό ξεκίνησε από το Μαρόκο. Πήγε στη Μαυριτανία, Σενεγάλη, Πράσινο Κροτήριο, Γινέα Βυζάου και όλη την δυτική εκτή της Αφρικής. Για τη διατήρηση των αποθεμάτων και για την βοήθεια προς τους αλείς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι αλείς πρώτοι και καλύτεροι ενδιαφέρονται για τη διατήρηση των αποθεμάτων. Κάποια άλλη κυρία εδώ με ρώτησε τι θα αλλάζαμε στη συμφωνία. Θα αλλάζαμε ότι βλέπουμε ότι δεν πάει καλά, ότι δεν λειτουργεί, ότι δεν φέρει αποτελέσματα. Είναι ξεκάθαρο, το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς με μια αναπτυσσόμενη χώρα είναι να την ε, καταρτήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει. Κατάρτιση. Οι περισσότεροι εδώ νομίζω ότι το καταλαβαίνει αυτό. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στις χώρες όπου μπορούμε να αλλιεύσουμε και τι γίνεται στις χώρες όπου δεν αλλιεύουμε πια. Όταν δεν υπάρχει έλεγχος, ρώτησε κάποιος για τον έλεγχο στην Μαυρετανία. Ε, τι γίνεται, άμα δεν υπάρχει έλεγχος, εμείς όμως αλλιεύουμε στα ύδατα μιας κυρίαρχης χώρας και ακολουθούμε τους νόμους της χώρας αυτής και όχι μόνο και αυτά που απαιτεί η δικιά μας η νομοθεσία και που έχουμε πετύχει να τα τηρούν οι στόλοι που αλλιεύουν στα συγκεκριμένα ύδατα. Το μέγεθος, ας πούμε, των δικτυών, η απόσταση από τις ακτές, οι περίοδοι αλίευσης, τα είδη, άμα βρίσκονται σε περίοδο μία αναπαραγωγής. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά και τα ξεχνάμε. Κάτι άλλο είχε να κάνει με αλείς στην Μαυριτανία που είπαμε ότι τους είδαμε χωρίς να φοράνε ε, ελέγχουν οι τοπικές αρχές τα πράγματα. Εμείς θέλουμε και στις περισσότερες περιπτώσεις το έχουμε πετύχει. Όπως έλεγε και η Ισπανίδα νωρίτερα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εμείς εκμεταλλευόμαστε τις θάλασσες. Πάνω από 30 χρόνια ασχολούμαι με την Αλία και η οικογένειά μου παλιότερα και ξέρουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τη θάλασσα. Έχουμε μεγαλώσει μαθαίνοντας ότι πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον όταν αλλιεύουμε. Αυτή την οτροπία πρέπει να καλλιεργήσουμε και στις τρίτες χώρες. Αλλιώς θα ζημιωθούμε. Η πολιτική μας πρέπει να πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να βοηθήσουμε τις τρίτες χώρες, αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε η οικονομία των χωρών αυτών δεν θα βελτιωθεί, δεν θα ενισχυθεί αν δεν ακολουθούν τους σωστούς κανόνες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα. Θα ήθελα να απαντήσω κυρίω στο ερώτημα εξή. Λέμε ότι τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο τη αμόρφωση τη κοινή ελευθερική πολιτική. Τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ νομίζω ότι αν κάνουμε κάτι πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας συνοχής για την ανάπτυξη. Υπάρχει μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε πριν από δύο χρόνια για τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη με ένα κεφάλαιο για την αλλία. Και στην τελευταία έκθεση του 2009 νομίζω υπογραμμίζονται πολλές ασυνάφειες. Και οι βασικές ε, είναι δύο ειδών. Και συμφωνούμε με αυτή τη διαπίστωση πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν ε, αμφιλεγόμενοι στόχοι όσον αφορά την εξωτερική διάσταση. Συγκρόναμε δηλαδή οι στόχοι. Και μερικέ φορές υπήρξε υπερδυναμικό στα ύδατα των τρίτων χωρών και δεν ε, έγιναν αρκετά στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε, δεν πρέπει αυτοί αυτές οι συμφωνίες να οδηγήσουν σε υπερβολική εργατικό δυναμικό ε, στις, ε, στα ίδια των δύο χωρών. Γι' αυτό θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις οικονομικές πτυχές από τις πτυχές που έχουν σχέση με την πρόσβαση στους πόρους και πρέπει αυτές οι εταιρικέ σχέσεις ε, να συμβάλλουν στη βελτίωση των, των επιπτώσεων επί του τοπικού παράγοντα. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε πάνω σε αυτά τα δύο πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη, στην τοπική ανάπτυξη. Όλα δεν είναι θέμα χρημάτων. Όπως έλεγε ένας Σενεγάλος ψαράς, δεν είναι με το να δίνει κανείς ε, χρήματα για τη φτώχεια ότι εξαλείφεται η φτώχεια. Δεν μπορεί ξαφνικά όλα αυτά τα χρήματα, 100-160 εκατομμύρια ε, ευρώ, με ένα μαγικό τρόπο θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Πρέπει να φροντίσουμε, να αντιμετωπίσουμε την... Να, να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν θα έχουμε αηφόρο ε, αλία, θα έχουμε διαφθορά. Τα χρήματα θα εξανεμιστούν δεν θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Θα δοθούν άδειε σε όποιον μπορεί να καταβάλει κάποιο τίμημα για αυτή την άδεια, χωρί διαφάνεια. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από πλευρά ανάπτυξη και να πούμε ότι χωρί μηχανισμό διαφάνεια και συμμετοχή δεν θα λειτουργήσει. Θα υπάρχει πάντα διαφθορά, θα υπάρχει πάντα έλλειψη συμμετοχή και τελικά δεν θα υπάρξει αηφόρο αλεία. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιος είπε ότι όλοι είναι κατά του ευρωπαϊκού ε, τομέα αλλιάς. Όχι, δεν συμφωνούμε. Αλλά θέλουμε να υποστηρίξουμε τον ευρωπαϊκό τομέα, διότι κατέδειξε ότι μπορεί να κάνει, επειδή μπορεί να κάνει αηφόρο αλλία και όχι επειδή ε, είναι ευρωπαϊκό τομέα. Πολλοί αλλοί από την Ευρώπη δεν ε, πραγματοποιούν αηφόρο αλλία. Μιλήσατε για την Κίνα δεν θέλω να κατανομάσουν μια χώρα, αλλά γεγονό είναι ότι η Κίνα έχει αρνητική επίπτωση ε, επί τη Αλία, κυρίω στη Δυτική Αφρική. Φυσικά λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε ώστε οτιδήποτε κάνουμε δεν θα οδηγεί σε μετατόπιση εμ, στόλων υπέρ των μη αηφόρων στόλων. Αλλά όλοι οι Ευρωπαίοι ε, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αηφόρο αλία. Οι περισσότεροι μπορούν, αλλά όχι όλοι ο κύριος Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ε, μην υπάρξει παρεξήγηση. Δεν είπα ότι ε, ορισμένοι δεν είχαν κανονισμός εάν η αλίες στη Μαυριτανία ε, υπάρχει αλία. Υπάρχουν άδειε για κάθε απόθεμα. Δεν είπα λοιπόν ότι ε, κυκλοφορούν χωρίς άδειε. Όχι. Δεύτερον, όταν μίλησα για πολλά πλοία στη θάλασσα, είπα αυτή είναι η ικανότητά τους, όποια και αν είναι. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Είναι μεγάλο το δυναμικό. Και η μόνη λύση, πιστεύω, είναι να εκφορτώνεται επιτόπου η παραγωγή επιτόπου, διότι είναι πιο εύκολο να ελέγχουμε ε, ε τα ψάρια επιτόπου. Διότι δεν μπορεί κανείς να τα ελέγχει όλα πάνω, εν πλώ. Δεν υπάρχει ένας στόλος επιτήρησης. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα που τέθηκε, για τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι το εξή. Ουσιαστικά, οι δύο πλευρές έχουν τα προβλήματά τους. Η Ευρώπη θέλει να γίνεται η αλία ώστε το πιο γρήγορα. Η Μαυριτανή και η Ευρωπαϊκή κυβέρνηση θέλει να έχει ορισμένα χρήματα το ταχύτερο δυνατόν. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Διότι λέμε ότι η οικονομική υποστήριξη γίνεται για την ανάπτυξη ε, του τομέα. Αλλά αφαίρετα δίνονται αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι ο προορισμό αυτό το κονδύλιο. Αν πούμε υπάρχουν 10 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση αηφόρου αελία στη Μαυριτανία, τι σημαίνει. Αν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, δεν θα χρηματοδοτηθεί σωστά. Εκτό εάν χρηματοδοτήσουμε τα υπάρχοντα προγράμματα. Και αυτό πάλι δεν γίνεται. Στη Μαυριτανία, για παράδειγμα, υπάρχουν τόσα εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν απορροφήθηκαν παρά το γεγονό ότι υπάρχει οικονομική υποστήριξη. Αλλά υπάρχουν βενθοπυλαγικά είδη και τα πλοία που είναι έτοιμα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ε, για αλία των μικρών μονάδων, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν αυτά τα προγράμματα και τα χρήματα είναι εκεί και δεν έχουν απορροφηθεί. Ένα άλλο στοιχείο. Όταν χρηματοδοτείται η έρευνα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και η επιτήρηση. Πολύ καλά. Αλλά αν προσθεθούν νέα πλοία, σε τι θα χρησιμεύσει αυτό. Εάν ε, υπάρχει ε, υπεραλία προς τι να γίνεται επιτήρηση. Θα επιτηρούνται μόνο τα παράνομα πλοία. Τα, λοιπόν, τα πλοία που με άδεια ε, αλλιεύουν θα υπάρξει υπεραλία τελικά. Γι' αυτό δεν θα υπάρχει πραγματική ανάπτυξη ούτε αηφόρος αλία. Θα πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα για την επιτήρηση, για την έρευνα χρηματοδοτείται η έρευνα από τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες χρηματοδότησαν αυτά τα δύο πλοία, ε, τα διερευνητικά πλοία στη Μαυριτανία. Και οι Γερμανοί μας έδωσαν χρήματα. Χρηματοδοτήθηκαν ε, από τους Γερμανούς. Και είπαμε υπάρχουν τέσσερα εκατομμύρια. Αλλά δεν βλέπω τα αποτελέσματα επιτόπου. Συνεπώς δεν υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα αυτών των αλληλευτικών συμφωνιών για την ανάπτυξη του λευτικού τομέα στη Μαυριτανία. Αυτά προσπάθησα να σας πω, ίσως τα είπα πολύ γρήγορα ε, στην ομιλία μου, αλλά τελικά θα ήθελα να πω το εξή. Νομίζω ότι η μόνη λύση για να προχωρήσουμε είναι τα ευρωπαϊκά πλοία να προσπαθήσουν να εγκατασταθούν σε αυτές τις χώρες, να δημιουργήσουν εργασίες γιατί τα υπόλοιπα είναι καπνός. Από τη δεκαετία του 70 παρακολουθώ τις ελευθερικές συμφωνίες και τίποτα δεν αλλάζει. Δεν μπορούν να αναπτυχθούν αυτές οι χώρες με βάση τις ελευθερικές συμφωνίες. Ε, οι, τα, χώρες που έχουν ε, πλοία μπορούν να αλλιεύουν, τίποτε άλλο. Δεν γίνονται επενδύσεις σε αυτές τις χώρες. Η Ισπανία είχε επενδύσει στη Μαυριτανία. Αλλά προτού υπάρξουν τα ισπανικά αλλιευτικά πλοία και κατόπιν ε, ε, εξέλιπαν αυτά τα πλοία. Εφόσον υπάρχει ο εξωτερικός στόλος που έχει την προτεραιότητα, δεν θα υπάρξει τοπική ανάπτυξη και δεν θα υπάρξει αηφόρος αλία, επειδή υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Ε, σας μίλησα για την Κίνα. Πράγματι, ε, δεν είπα ότι η Κίνα παρενέβη για να πάρει τη θέση των Ευρωπαίων. Όχι, είπα ότι η Κίνα παρενέβη επιδέξια χρηματοδοτώντας ένα τοπικό στόλο που είχε, ήταν πεπαλαιωμένος και χρηματοδότησε την ανανέωση του στόλου η Κίνα. Και είπα πάλι ότι υπάρχουν δυνατότητες μέσω της χρηματοδότησης προστιθέμενης αξίας των μεταποιημένων προϊόντων στη Μαυριτανία. Και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Μορφή συνεργασία. Ίσως θα πρέπει να αλλάξει η μορφή τη συνεργασία μας για να καταλήξουμε σε μία λύση. Να υπάρξουν επενδύσει περισσότερες επί τόπου, όχι σε χρήματα. Σημαντικό είναι, δεν είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικό είναι η παρουσία και η δημιουργία θέσεων εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πολύ σημαντικές διευκρινήσεις. Το λόγο έχει η κυρία Φίσκνες. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που διατυπώθηκαν. Μία ήταν τι δίνει η Νορβηγία όσον αφορά την αλία για την ε, συνεργασία και την ανάπτυξη είναι περίπου 20 έως 25 εκατομμυρία ευρώ ετήσια αυτό το ποσό. Επίσης με ρωτήσατε, να, μου ζητήσατε να σχολιάσω σε σχέση με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να κάνει, τι να πράξει. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, να δώσω κάποιες συστάσεις. Μακροπρόθεσμα νομίζω, μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση και η διαφάνεια είναι κέρια σημασία στοιχεία. Όμως και ανέφερα Επίσης, τι φάνηκε να είναι καλό, θετικό με την βοήθεια για την ανάπτυξη που προσφέρει η Νορβηγία. Δεν θα ήθελα όμως να υποβάλω συστάσεις προς την ΕΕ. Τώρα, αξιολογήσεις αποθεμάτων και Βορειοδυτική Αφρική και μέσω του προγράμματος Νάνσεν υπάρχει υποστήριξη επίσης για την χρήση των τοπικών αυτών δυνατοτήτων σκαφών για τέτοια αξιολόγηση αποθεμάτων. Και έχει η Μαυριτανία αυτή τη δυνατότητα, αυτό το σκάφο το ερευνητικό, το οποίο χρησιμοποιείται για έρευνε για την αξιολόγηση αποθεμάτων. Αν τα στοιχεία από το πρόγραμμα Νάνσεν ή από το, στοιχεί, από το σκάφος αυτό, αν επαρκούν για να μπορέσει κανείς να τοποθετηθεί για την κατάσταση των αποθεμάτων, δεν το γνωρίζω. Όμως θα ήταν περίεργο αν δεν θα μπορούσε κανείς να πει τίποτα με αυτά τα στοιχεία. Διότι εδώ και 20 χρόνια υπάρχει προσπάθεια συλλογής στοιχείων και αξιολόγησης φυσικά και με τα κράτη στη Βορειοδυτική Αφρική αυτών των αποθεμάτων, αυτών των πόρων. Έτσι λοιπόν θα λέγα ότι υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Τώρα από την άλλη πλευρά θα έλεγα ίσως ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να υφίσταται με συμφωνίες ε, είναι ότι μπορεί να υπάρχουν δύο συμφέροντα τα οποία θα είναι δύσκολο να διαχωριστούν το ένα από το άλλο. Ο τομέας των κρατικών συμφερόντων είναι η μία πλευρά. Όταν εργαζόμαστε στην βοήθεια για την ανάπτυξη, είναι πραγματικά το συμφέρον των αναπτυσσομένων χωρών στο οποίο επικεντρωνόμαστε. Και αν συγχαίει κανείς αυτές τις δύο πλευρές, αυτές τις δύο όψεις του νομίσματος, δεν θα είναι τόσο εύκολο να διαπιστώσει τι είναι εκείνο το οποίο επιθυμεί κανείς. Τα δικά του συμφέροντα εξυπηρετεί δηλαδή κανείς ή τα συμφέροντα της αναπτυσσόμενης χώρας. Τι γίνεται. Και η διαφάνεια εδώ και ο ανοιχτό χαρακτήρας του εγχειρήματο είναι κέρια σημασία στοιχεία διατρέχοντας αυτό το εγχείρημα συνολικά. Αυτά ήθελα να πω και νομίζω απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πρόεδρο σας, ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Διευθυντή. Μιλάτε παρακαλώ. Λυπούμε πολύ που ε, αναγκαστήκατε να ε, χάσετε την ευκαιρία. Παρακαλώ. Merci, merci pour ces... Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργάνωσε τη συνάντηση αυτή, στην οποία προσκάλεσε και μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει την μεταρρύθμιση της κοινή ελληνικής πολιτικής, την διάσταση την εξωτερική ιδιαίτερα και κυρίως τις αλλιευτικές συμφωνίες. Εδώ και αρκετούς μήνες τώρα οργανώνουμε συναντήσεις με κάθε πλευρά, με όλους τους φορείς Πολλοί από αυτούς μάλιστα μίλησαν εδώ σήμερα. Η συνάντηση αυτή μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας συγνώμη καταρχήν για το μπέρδεμα που έγινε και δεν ήρθε ο πυρογνώμονας ο οποίος έπρεπε να έρθει και να πάρει το λόγο εδώ όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Ζολή. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εμπειρογνώμων είναι στη διάθεσή σας, άπαξ και θέλετε να του ζητήσετε να έρθει, είναι στη διάθεσή σας. Δεύτερο ζήτημα που ακούσαμε στην αρχή της συνεδρίασης, αν δεν απατώμε, δεν είχα έρθει ακόμα, αλλά ήταν το εξής. Τι δίνουμε στις νήσους Σόλομον. Στα νησιά του Σολομόντα. Έχουμε τρεις συμφωνίες με τον Ειρηνικό, με τα νησιά του Σολομόντα, με την Μικρονησία και με το Κυριμπατή. Είναι τρεις συμφωνίες μικρές όσον αφορά τα κονδύλια, γιατί είναι μικρές και δυνατότητες αλίευσης που υπάρχουν για τα ευρωπαϊκά σκάφη στις ζώνες αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης. 65 ευρώ, ακούσατε σήμερα το πρωί, αυτό το ποσό έχει να κάνει με την κατανομή του βάρους ανάμεσα στο κοινοτικό προϋπολογισμό και τους πλειοκτήτες. Είναι δηλαδή κατανομή που βασίζεται στην αξιολόγηση 100 ευρώ τόνος τόνου που είναι σημείο αναφορά και χρησιμοποιείται για όλε τι συμφωνίε που έχουν να κάνουν με τον τόνο. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή με τι νήσου του Σολομόντα. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται και στις άλλες συμφωνίες για τον τόνο. Τώρα, στα νησιά του Σολομόντα υπάρχουν τέσσερα ε, σκάφη με γρίπο. Δεν υπάρχουν ε, παραγαδιάρικα. 10 ή 12 στις άλλες συμφωνίες ε, σκάφη με γρίπο το ποσό της άδεια αλίας για τις νήσους Σολομόντος είναι 20.000 ευρώ. Και για να καταλάβετε, στις Σεχέλε σήμερα η άδεια είναι 61.000 ευρώ. Και οι σεχέλε είναι ένα μέρος όπου τα τονοθερικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλά και ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής το παίρνουμε, υπάρχει ένα κύκλωμα ε, μεγάλο. Τώρα κάποιος από σας θέλει περισσότερες διευκρινήσεις όσον αφορά τα οικονομικά αυτά στοιχεία, είμαστε εννοείται στη διάθεσή σας. Γραπτά μπορούμε να σας τα δώσουμε, αλλά δεν θα έπρεπε τώρα να αρχίσω να σας βομβαρδίζω με νούμερα. Θέλω να πάω πάλι λίγο σε κάτι που είπε η κυρία Ζολή πριν και έχει δίκιο. Ότι οι ελευτικές συμφωνίες δεν είναι συμφωνίες για την ανάπτυξη. Και στο κάτω-κάτω ποτέ δεν είπαμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για οικονομικές συμφωνίες που έχουν όμως μία αναπτυξιακή πτυχή. Εξάλλου, αυτό φαίνεται και από τα ποσά. Γιατί δεν προέρχονται από την αναπτυξιακή πολιτική, αλλά από έναν ιδιαίτερο προϋπολογισμό που είναι ακριβώς οι ελευτικές συμφωνίες. Όμως, παρά το γεγονός ότι τα ποσά είναι λίγα, γιατί μιλάμε για 166 εκατομμύρια το χρόνο συνολικά και ένα μέρος μόνο πάει στην ανάπτυξη, επειδή έχω αρκετά χρόνια που ασχολούμαι με την ανάπτυξη, θα έλεγα ότι με τα ποσά αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας κάνουμε ανάπτυξη. Και άκουσα κάποιον από τους συμμετέχοντες που είπε ότι θα ήταν καλό να κάνουμε έναν απολογισμό σε βάθος τι γίνεται με την ανάπτυξη. Η προσθεθέμενη αξία νομίζω ανά ευρώ σίγουρα είναι κάτι πιο θετικό από άλλα ευρώ που ένα εκατομμύριο πάνε σε άλλους τομείς. Αυτού του είδους η συνεργασία βασίζεται στην παρουσία επαγγελματιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτόπου και μας επιτρέπει να έχουμε συνεργασία όπου συμμετέχει, που συμμετέχουν και οι δημόσιες αρχές, αλλά υπάρχει και συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου. Υπάρχουν επενδύσεις που γίνονται στις χώρες. Υπάρχει μεταφορά τεχνολογίας επίσης. Υπάρχουν ε, ε, ναυτικοί οι οποίοι μεταφέρονται με τα σκάφη αυτά. Τέλο πάντων ο απολογισμός δεν είναι τόσο αρνητικός όπως περιγράφηκε. Φυσικά μέσα στα πλαίσια των ελάχιστων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας για να φροντίσουμε για την ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα εξάλλου μετρούνται με τον έλεγχο και την εποπτεία συνολικά. Και βάση της διαφάνειας. Να, ένα πολύ βασικό στοιχείο. Η δραστηριότητα των Ευρωπαίων αλλιέων διέπεται από διαφάνεια. Και ακριβώς επειδή υπάρχει διαφάνεια, γι' αυτό και αποτελούν έναν εύκολο στόχο όποιου θέλει να επικρίνει. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν αγνοούμε τώρα που προετοιμάζουμε τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής ε, πολιτικής, τα έχουμε εντοπίσει. Και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει πολύ σύντομα στις συμφωνίες αυτές να εισαγάγει μια ρήτρα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατικές αρχές, που στο κάτω-κάτω είναι εκείνος τόπος για τις άλλες ευρωπαϊκές συμφωνίες. Και έτσι, χωρίς να έχουμε νομικές δυσκολίες, μπορούμε να σταματήσουμε αυτές τις συμφωνίες αν δεν τηρούνται οι ρήτρε αυτές. Ενώ τώρα δεν μπορούμε. Επίσης, μια ρήτρα κατά της διαφθοράς πιστεύουμε ότι είναι ευπρόσδεκτη σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Ένα άλλο στοιχείο στις συμφωνίες αυτές είναι μια ρήτρα διαφάνειας που έχει να κάνει με την χώρα εταίρο. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι κάνει αυτή η χώρα εταίρος με τους Κινέζους ή με δεν ξέρω ποιους άλλους για ένα πολύ απλό λόγο. Βάσει του διεθνούς δικαίου δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε λευτική συμφωνία παρά μόνο στο περισεβούμενο από τους πόρους. Ενώ αν δεν γνωρίζουμε τι κάνει το συγκεκριμένο κράτος που αποφελείται από τις συμφωνίες μας αυτές με το πλεόνασμα των πόρων του, μπορούμε πάντα να χρηματοδοτήσουμε επιστημονική επιτροπή, να κάνουμε αξιολόγηση των αποθεμάτων, αλλά ποτέ δεν θα είμαστε σίγουροι για το τι χρησιμοποιούμε εμείς αν χρησιμοποιούμε όντω το πλεόνασμα ή όχι. Ένα λοιπόν από τα μεγάλα θέματα των νέων συμφωνιών θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της επιστημονικής πτυχής έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται με το πλεόνασμα. Αν μη τι άλλο γιατί έχουμε την υποχρέωση αυτή βάση του εφαρμόσιμου διεθνούς δικαίου. Εδώ θέλω επίσης να αναφέρω και ένα άλλο πρόβλημα που είναι της έλλειψης ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες ανάπτυξης μιας χώρας και των ποσών που μπορούμε εμείς να κινητοποιήσουμε. Όπως έλεγα και πριν, πρόκειται για οικονομικές συμφωνίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την αξία μιας συμφωνίας εξαρτάται από τις δυνατότητες αλίευσης που υπάρχουν. Αποτέλεσμα, είναι αλήθεια ότι στον Κυριμπατή, για παράδειγμα, ή στις νήσους του Σολομόντα έχουμε συμφωνίες ποσών που δεν επαρκούν. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός. Οι υπολογισμοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πολύ πιο αυτόνομα τις αναπτυξιακές ανάγκες των χωρών εταίρων. Μερικές φορές δεν φτάνουν τα ποσά, άλλες φορές είναι παραπάνω πόσα χρειάζονται για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, τα ακούσαμε με την ε, αξιολόγηση σήμερα υπάρχουν λόγοι που δεν έχουν άμεση σχέση με την αλία μερικές φορές, αλλά έμεση. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την αξιολόγηση των συμφωνιών αυτών. Αυτά, αυτό εδώ ισχύει και για την Βερλανδία, όπως όλοι ξέρουμε. Θέλω επίσης να αναφερθώ λιγάκι και σε κάτι άλλο προς ενημέρωση της εμπειρογνώμονος που έχουμε από την Νορβηγία. Ότι και η Νορβηγία υποφελείται από ελευτικές συμφωνίες, ακόμα και αν αυτό γίνεται έμεσα. Έχουμε κάποιες ανταλλαγές με την Νορβηγία. Η Νορβηγία αλλιεύει χάρη σε αυτές τις αλλιευτικές συμφωνίες. Συνεπώς, πρέπει να διορθωθούν τα προβλήματα και να υπάρχει λογική με την αναπτυξιακή πολιτική. Να υπάρχει μια σχέση πολύ πιο σοβαρή από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Και δύο πλευρές πρέπει να παίξουν πάντως αυτό το παιχνίδι. Και κυρίως εδώ θα αναφέρω μία πτυχή που είναι η προπτική μιας περιφερειακής προσέγγισης όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία. Υπάρχουν διαφωνίες εμείς δεν πιστεύουμε ότι η διακυβέρνηση μπορεί να οργανωθεί σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί πρόκειται για το κράτος δικαίου. Και το κράτος δικαίου είναι μέσα σε χώρες σήμερα και όχι περιφερειακά. Περιφερειακά μπορούμε να λέμε πολύ ωραία λόγια, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια πραγματικά χρηστή διακυβέρνηση της Αλίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε διακυβέρνηση σε περιφερειακό επίπεδο. Ό,τι προτάσει προτάσεις συγκεκριμένες έχετε, εφικτές να τις συζητήσουμε. Πάντως σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει και το έχουμε αποδείξει στον ειδικό ωκεανό η δυνατότητα για συνεργασία ακόμα και με περιορισμένα κονδύλια ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου. Δύο λεπτά ακόμα μπορώ. Ρωτάει ο μιλητής. Πολύ σύντομα για τα σχόλια τα οποία ακούσαμε. Συμφωνώ με την κυρία Λόβιν λέγοντας ότι οι στόχοι που ορίστηκαν πριν από 10 χρόνια για την κοινή ελευθερική πολιτική και την εξωτερική διάσταση πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν. Σίγουρα συμφωνώ λέγοντας ότι η πρόθεση της αηφόρου αλίας είναι ένας ουσιαστικός στόχος για την εξωτερική διάσταση επειδή είναι μια σημαντική διάσταση τη εσωτερική διάσταση και λοιπόν θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο εξωτερικό. Δεύτερο στόχο για μα είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για να πλαισιώσει τη δραστηριότητα ε, της, του στόλου μας σε μακρινά ύδατα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να καταλήξουν στην καταστροφή αυτού του πλαισίου. Οτιδήποτε συμβάλλει στην καταστροφή του πλαισίου διακυβέρνησης πρέπει να εξαλειφθεί. Να υπάρξει πλήρη διαχωρισμός τώρα μεταξύ συνεργασίας στην ανάπτυξη και την αλία με τρόπο καθόλου συνδεδεμένο με τον Ευρωπαϊκό Στόλο και με τη συνεργασία ε, στα πλαίσια του Στόλου της Ευρώπης, πιστεύω ότι προσκρούει σε ορισμένε αλήθειες που θα την θυμίσω. Στον τρόπο με τον οποίο σήμερα διαμορφώνουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με βάση τη συμβολή των χωρών εταίρων και των προτεραιοτήτων ανατομέα, κανένας δεν έχει καθορίσει ότι ο τομέας ελίας είναι προτεραιότητα στην ανάπτυξη. Δεύτερον, ε, το οικονομικό σκέλος, εξελίφουμε και την ύπαρξη ε, ανάπτυξη από πλευράς ε, μεταφοράς τεχνολογίας και επενδύσεων και η πολιτική ανάπτυξη γίνεται μια πολιτική που θελοποιείται μόνο από συμβούλους, ζητώ συγγνώμη στους συμβούλους, τους οποίους σέβομαι πολύ. Τώρα, για την αξία των εκφορτώσεων. Μπορώ να σας δώσω προσώτες λεπτομέρειες. 443 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά μέσον όρο. Αλλά αυτό είναι ένας γενικός αριθμός. Ε, μπορεί τα ψάρια να εκφορτωθούν στην Ευρώπη ή στην Αφρική. Ένα μεγάλο ποσοστό ε, των ελευμάτων από τα πελαγικά πηγαίνουν στην Αφρική και πολλούνται ας πούμε στην αγορά της Νιγηρίας ή εκφορτώνονται σε άλλες χώρες, Νότια Αμερική, όπου υπάρχουν τα δίκτυα για την μεταποίηση των ηχθείων. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στο δικό σας το ερώτημα για τη Γρυλανδία. Ο λόγος της υποχρησιμοποίησης των δυνατοτήτων αλληλείας με τη Γρυλανδία είναι ότι αυτές οι αλληλευτικές δυνατότητες υπολογίστηκαν μεν, αλλά είναι φανερό ότι κάθε χρόνο γίνεται επιστημονική αξιολόγηση αυτών των ηλεκτρικών δυνατοτήτων και παρέχονται ε, στον Ευρωπαϊκό Στόλο και στους άλλους στόλους μόνον όσα επιστημονικά είναι αποδεκτά. Συνεπώς, βλέπουμε ότι οι ελευτικές δυνατότητες δεν χρησιμοποιούνται όλες και καθόλου στα πλαίσια της συμφωνίας με τη Γρυλανδία. Και μάλιστα, αυτή είναι μια συμφωνία η οποία θα αναθεωρηθεί. Θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Άλλοι θέλουν να παρέμβουν, όπως πρέπει να τερματίσουν και οι διερμηνείς με την εργασία τους. Θα δώσω τον λόγο συνέχεια στην κυρία Ζολή. Ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ την κυρία Ζολή βέβαια, είναι αυτονόητο. Και όλου τους Ευρωβουλευτές τη Επιτροπή Ανάπτυξη για την παρουσία τους εδώ και την κοινή συζήτηση αυτών των θεμάτων που ήταν ενδιαφέρουσα νομίζω και ήταν επωφελήσα για αμφότερες πλευρές. Ε, και ένα λεπτό ακόμα. μα έδωσαν πέντε λεπτά οι διερμηνεί. Ε, Λέω ότι θα ολοκληρώσουμε σε ένα λεπτό. Θα λάβει τον λόγο η κυρία Ζολή μετά λίγη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους μίλησαν για τη συμβολή τους, την πολύ σημαντική συμβολή και ε, πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να επαναπροσδιορίσουμε ένα μέρος αυτών των αλληλευτικών συμφωνιών να λάβουμε υπόψη το ότι η εποχή όπου ο Ευρωπαϊκός Στόλος μπορούσε να μην τηρεί τους κανόνες, έχει παρέλθει, όπως και πολλά άλλα πράγματα, υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη αυτή τη στιγμή, μια δυναμική και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε το 2011 το 2010 να κάνουμε όσα κάναμε πριν από 10 ή 20 χρόνια. Το ζητούμενο είναι διαφορετικό. Συνεπώς, θα πρέπει να αναμορφωθεί η ε, σύμβαση των εταιρικών σχέσεων με την Αλία, λαμβάνοντας υπόψη ε, τα νέα δεδομένα όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση, την αηφόρο Αλία και επίσης όσον αφορά την κατανομή των πόρων και τη δίκαιη κατανομή μεταξύ των παρακτήων χωρών, όλα αυτά θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Αλλά νομίζω